good morning um, well. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην δημόσια αυτή ακρόαση με θέμα πέραν της μείωσης ε, ε, των αερίων του θερμοκηπίου και των, uh, του του άνθρακα, της διαρρής διοξιδίου του άνθρακα από το 20% Έχουμε το πάνελ προσκεκλημένο και τον κύριο Ματία Κόρτ που είναι μέλος της ομάδας εργασίας για το θέμα αυτό, για τις μείωσεις πέραν του 20%. Έχουμε και τον κύριο Μπάσεκ Χάουτ που ασχολείται με το ίδιο θέμα και κανονικά θα πρέπει να έχουμε μαζί μας και κάποιον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μαρή Ντόνελη από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας αλλά δυστυχώ η Μαρή δεν έχει έρθει ακόμη. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταφτάσει και εκείνη. Θα ήθελα στα εισαγωγικά σχόλια να σας υπενθυμίσω ότι εννέα μήνες πριν την επόμενη διάσκεψη κορυφής για το κλίμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπαθεί να αποκρισταλώσει τη γνώμη της. Και από τότε που έχουμε υιοθετήσει τη μονομερή μας δέσμευση το Μάρτιο του 2007 για να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου για 20, κατά 20% πολλά έχουν αλλάξει. Για να μην μιλήσουμε για τα τελευταία γεγονότα στην Ιαπωνία. Αλλά ας μείνουμε στο περιεχόμενο, ας περιοριστούμε στο περιεχόμενο της δημόσιας αυτής ακρόασης και να μην ενδώσουμε στον πειρασμό να επεκταθούμε στις εξελίξεις στην Ιαπωνία. Ας περιοριστούμε λοιπόν στο σημερινό μας αντικείμενο και να πούμε ότι και άλλοι εταίροι μας έχουν προβεί σε περιορισμούς και έχουν δεσμευτεί να μειώσουν την θέρμανση του πλανήτη σε δύο, κατά δύο βαθμούς και μάλιστα οι τεχνολογίες με χαμηλή χρήση άνθρακα αρχίζουν και γίνονται ανταγωνιστικές, είναι αναμφίβολο. Οπότε με όλες αυτές τις εξελίξεις ε, διερωτόμαστε μήπως δικαιολογούνται περαιτέρω μονομερείς δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο του Μαρτίου του 2007 συμφώνησε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, να φτάσουμε στο 30% αν και όλες οι υπόλοιπες περιοχές του κόσμου ε, υιοθετήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Η έκθεση αυτή που είναι η βάση της σημερινής δημόσιας ακρόασης και λέει για μείωση των ε, εκπομπών πέραν του 20% του κυρίου Eckhout Και ε, έχουμε και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Ήτρε της κυρίας Γιόρνταν Σίζελ, δυστυχώς απουσιάζει. Θα πρέπει με αυτήν την έκθεση αυτή να ευκρινίσουμε αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τι μέσα και μηχανισμούς έχουμε για να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου πέραν του 20%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει και έναν οδικό χάρτη για περιορισμό της χρυσά μέχρι το 2050. Έχουμε και το σχέδιο ενεργειακής αποδοτικότητας που υπέβαλε ο Επιτροπό Έτιγκερ. Και τα δύο αυτά έγγραφα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα θα αποτελέσει κλειδί για την υλοποίηση των τωρινών μας στόχων αλλά και των πιο φιλόδοξων στόχων, πέρα του 20% δηλαδή μείωση. Γι' αυτό προσκαλέσαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξετάσουμε τις τελευταίες της προτάσεις για τον τομέα αυτό. Θα ήθελα επίσης μια και απουσιάζει η Ρωμάνα Τζόρνταν, η συγκεντρια της Ήτρα, να αναφερθώ σε ορισμένα σύντομα ε, ζητήματα που περιέλαβε στην γνωμοδότησή της, της Επιτροπής Ήτρα. Καταρχήν, ε, η Ρωμάνα δίνει έμφαση και χαιρετίζουμε όλη αυτή την έμφαση σε μακροπρόθεσμες πολιτικές και όχι μόνο στον περιορισμό των στόχων της στρατηγικής του 2020. Επίσης, διευκρινίζει ότι η περαιτέρω μείωση των εκπομπών πέραν της του συμφωνημένου στόχου του 20% θα πρέπει να συνοδευτεί από τα κατάλληλα ενάψματα και όχι από συμπληρωματικά νομοθετικά μέτρα. Κατά συνέπεια, το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να θεσπίσει τις σωστές προτεραιότητες και να αφιερώσει περισσότερα κονδύλια σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και ενοτομία και να δώσει ενάψματα για τη χρήση, για την αξιοποίηση των κονδυλίων για μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας. Παράδειγμα, ανακαίνιση των κτηρίων κτλ. Αυτές είναι οι εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις. Αναφερθήκαμε στα βασικά στοιχεία της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ήτρε και χωρίς άλλη καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ματίας Γκρότ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα από πλευρά μου επίσης. Σήμερα έχουμε ένα σημαντικό θέμα στη μέση διάταξη. Πώς θα διαμορφώσει την κλιματική της πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Το 2008 εγκρίναμε ένα ευρύτατο πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια και είναι ακόμα επίκαιρο. 20% μείωση του οξυδίου του άνθρακα αποφασίστηκε και αν άλλοι μεγάλοι οικονομικοί εταίροι και συνασπισμοί ε, μας ακολουθήσουν, είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε μέχρι και το 30% στη μείωση σκέψεις έγιναν για το κλίμα και στην Κοπεχάγη και στην Κανκούν και είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι διεθνώ δεν υπάρχει πολύ μεγάλη προθυμία προ την κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα μεσολάβησε και η κρίση οικονομική και χρηματοπιστωτική, οπότε και η βιομηχανία και η οικονομία επλήγησαν. Σιγά σιγά επιστρέφουμε σε επίπεδα ομαλότητας, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί όμως η ανάκαμψη. Την περασμένη εβδομάδα μας ήρθε και αυτή η είδηση της Ιαπωνίας. Τρεις είναι οι θεομηνίες, τρεις είναι και οι καταστροφές, όχι μόνο θεομηνίες. Και υπάρχει κόσμος που λέει ότι εγώ δεν θέλω να το ζήσω αυτό στην Ευρώπη, αυτή την άλλη συνδοτή αντίδραση. Ε, ωστόσο και τα γεγονότα στην Ιαπωνία θα επηρεάσουν τη μελλοντική συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε τον Επίτροπο εχθέ και προχθέ στις διάφορες επιτροπές και αντέδρασε αμέσω και μάλιστα με τρόπο πάρα πολύ ταχύ και ε, ορθό και ανέλησε για αναλύει αυτό τον καιρό με τι υπηρεσίε του τι πρέπει να κάνουμε τους επόμενους μήνες και τα επόμενα έτη. Τι έχει σημασία τώρα σήμερα στην ακρόαση. Να συνενοηθούμε με ε, τους επιστήμονες ε, να δούμε τι επιπτώσεις έχει το λεγόμενο carbon leakage, δηλαδή ότι σηκώνονται και φεύγουν οι επιχειρήσεις που παράγουν διοξίδιο του άνθρακα. Εμείς ανταγωνιζόμαστε διεθνώς ως βιομηχανία και αν η Ευρώπη έχει μονομερείς κανόνες και μάλιστα πολύ πιο αυστηρούς, πρέπει να δούμε πώς αυτό επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. αν έχουμε πιο αυστηρή νομοθεσία για το περιβάλλον, αυτό έχει επίδραση εκτός από τη δική μας ανταγωνιστικότητα και σε κάποιους εταίρους. Τους επηρεάζουμε, δεν τους επηρεάζουμε, δεν έχει κανένα νόημα ή η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Σε ποιους τομείς μπορεί άρα η Ευρώπη να προχωρήσει χωρίς να πλήξει την ανταγωνιστικότητά της. Έχει νόημα να το κάνει. Ποιοι οι στόχοι είναι αυτοί, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προς τα πάνω, 40% π.χ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τεχνικά υπάρχει δυνατότητα θεωρητικά, αλλά οι συνέπειες ποιες θα είναι στο συνολικό οικοδόμημα της οικονομίας. Και επίσης θα πρέπει να δούμε και το οικολογικό στοιχείο. Αν η Ευρώπη μονομερός προχωρήσει περισσότερο, θα υπάρχουν οικολογικές συνέπειες. Και ποιες είναι αυτές. Επηρεάζει τίποτα και σε ποιο βαθμό αυτό. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε, να τα διαπιστώσουμε και στο τέλος αυτής της προσπάθειας, τον Ιούνιο, ο κύριος Χάουτ έχει το χρονοδιάγραμμα στο μυαλό του, θα εγκρίνουμε μια έκθεση πρωτοβουλία. Το είπαμε και χθε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μπορεί να συγκρουστούμε ε, και στην ψηφοφορία, αλλά σε μια έκθεση πρωτοβουλία δεν νομίζω ότι έχει νόημα να πάμε διχασμένοι στην ψηφοφορία. Γιατί είναι που είναι έκθεση πρωτοβουλία, αν δεν είμαστε και ενωμένη δεν θα πιάσει τόπο και δεν θα περάσουμε καθόλου τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Έχει λοιπόν καθήκον το Κοινοβούλιο να δει και την πλευρά του περιβάλλοντος, αλλά να ακούσει και τα επιχειρήματα της οικονομίας, της βιομηχανίας και της ανταγωνιστικότητας και να τα αναλύσει ε, όσο και να τα συνδυάσει. Γι' αυτό είναι μια κριτική που ακούμε και στο Κοινοβούλιο. Και βλέπω το συνάδελφο Ρομπέρ Γκέβελ. Το έχουμε συζητήσει. Από το 2008 το συζητούσαμε για το πακέτο ε, για την ενέργεια και το εγκρίναμε, το κλίμα μάλλον, σε πρώτη ανάγνωση. Το Κοινοβούλιο επέμενε και σωστά. Αλλά αυτό άφησε πικρή γεύση σε πολλούς συναδέλφους και θα πρέπει τώρα να μπούμε στο κόπο να κάνουμε αναλύσεις ε, πάρα πολύ ακριβείς, πάρα πολύ σωστές, γιατί εμείς θα χρειαστεί να το υπερασπίσουμε αυτό, αν πάρουμε απόφαση ε, στα κράτη μας, στον κόσμο μας και να μην λέει κάποιος ότι ε, εμείς το πετύχαμε και κάποιοι άλλοι να λένε οι άλλοι φταίνε. Όχι, το Κοινοβούλιο ολόκληρο είναι πίσω από την προσπάθεια. Και θα χρειαστεί ακριβώς χρόνος για την ανάλυση αυτή. Χαίρομαι που έχουμε σήμερα εδώ εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη για να μας ενημερώσουν για το hearing, την ακρόασή μας. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Ελπίζω να είναι χρήσιμη και καρποφόρα η σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Μπάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πιλάρ. Λέγομαι Μπάς Εκχάουτ και είμαι η ε, εισηγητής Επιτροπής Περιβάλλοντος και μετά αυτή τη ακρόαση που είχαμε στην Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος και τώρα εδώ στην Επιτροπή Βιομηχανίας με τη Γιορτάνα ε, βλέπουμε ότι αυτό το θέμα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό. Είναι όλο και περισσότερο και βιομηχανικό. Καλό είναι λοιπόν, εκτό από την Επιτροπή περιβάλλοντο να τα εξετάζει αυτά και η Επιτροπή ε, που ασχολείται με την ενέργεια και τη βιομηχανία, για να ακούμε και τα δύο επιχειρήματα και να δούμε πώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Η έκθεση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αρχίζει από ένα σχέδιο και θα πρέπει να συνεννοηθούμε και με την εισηγήτρια τη Ρωμάνα Τζόρνταν Σίσελη της Επιτροπής εδώ Ήτρε και θα πρέπει να είμαστε και φιλόδοξοι. Πέρσι το Μάιο ήδη έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συστάσεις τη και είπαν ότι αν θέλουμε να έχουμε ε, μια λογική σχέση κόστους ωφέλειας, το 20% μέχρι το 2020 δεν φτάνει. Εγώ το μετέφρασα αυτό στην εκθεσή μου σε 30% μονομερής ε, μείωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το ακούμε από όλα τα επιστημονικά δεδομένα και επιχειρήματα. Από την πλευρά του κλίματος είναι σαφές το ότι αν θέλουμε να έχουμε διπλό στόχο και να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε 30% είναι ένα μόνο βήμα Αρχές Μαρτίου ε, ξεκίνησαν αυτά. Αν θέλουμε λοιπόν μέχρι το 2050 να είμαστε αποτελεσματικοί και ως προς το κόστος και την ωφέλεια πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τούτη εδώ την Επιτροπή. Δεν είναι μόνο το περιβαλλοντικό ε, επιχείρημα. Ας δούμε τι λέει η οικονομία, τι λέει η βιομηχανία, τι λέει η ανταγωνιστικότητα και η ενέργεια. Και ένα από τα επιχειρήματα κλειδιά είναι, αν δούμε την οικονομία μας, αν περάσουμε από το 20% στο 30% αυτό θα σημαίνει 40 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερες εισαγωγές πετρελαίου. 40 δις. Και αυτό έχει υπολογιστεί με μια τιμή βαρελιού στα 88 δολάρια. Γνωρίζουμε ότι τώρα είναι πολύ περισσότερο από 100 και η τάση οδική τη τιμής του πετρελαίου. Όσο πιο ακριβό είναι το πετρέλαιο λοιπόν, τόσο περισσότερα χρήματα θα εξοικονομήσουμε αν μειώσουμε τις εισαγωγές μας και αν αυξήσουμε τους στόχους για το κλίμα. Υπάρχουν πολύ σημαντικά στοιχεία. Είναι το τομέα ETS και μη ETS, ε, τις συναλλαγές ε, των δικαιωμάτων εκπομπών. Και χαίρομαι που θα το συζητήσουμε και εδώ, και την έρευνα και την ανάπτυξη και την καινοτομία. Θα πρέπει και οι αγορές να ανταποκριθούν και η οικονομία, αλλά εάν δεν κάνουμε τις απαραίτητες επενδύσεις, δεν, δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα. Δεν θα είναι ισορροπημένη εννοώ η πολιτική μας. Γι' αυτό θα ε, χρειαστεί να ε, το μελετήσουμε. Από την άλλη, εξοικονόμηση ενέργειας. Αν διαβάσετε τον οδικό χάρτη, αυτό το roadmap της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, τι λέει. Εάν φτάσουμε στο στόχο του 20% για το 2020, ήδη είμαστε στο 25% ε, των μειώσεων των εκπομπών. Έχουμε ξεπεράσει ήδη το 20% αν ε, καλύψουμε τους άλλους στόχους για εξοικονόμηση ενέργειας και για τις ανανεώσιμες. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα γίνει αυτό. Στο Κοινοβούλιο η συντριπτική πλειοψηφία ζητάει στόχους δεσμευτικούς. Και το ζήτησε ο Μπεν Μπένσεν στην έκθεσή του, με στόχους για εξοικονόμηση ενέργειας. Αν διαβάσετε όμως το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά, δεν είναι δεσμευτικά ακόμα τα μέτρα. Και χαίρομαι που είναι βασικό στοιχείο της ατζέντα και αυτό. Πώς θα βεβαιωθούμε ότι εξοικονομούμε ενέργεια και ότι αξιοποιούμε και το δυναμικό από αυτό που υπάρχει. Να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας, η αποδοτικότητα είναι κομβική. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ πάρα πολύ με τον Ματίας Γκρότερ Τελικά δεν θέλουμε να συγκρουστούμε στη ψηφοφορία 50 υπέρ 50 κατά με τοπικά. Θα πρέπει να φτάσουμε στους στόχους μας λοιπόν και ε, ε, σε άλλους στόχους από το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουν εμπόριο χωρίς μεταξύ τους για τα δικαιώματα. Αυτό που θέλουμε μειώνουν την εκπομπή ε, αερίων. Θα πρέπει ε, όμως να ε, προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας για την ενεργειακή απόδοση. Εμείς ως Κοινοβούλιο μπορούμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις πιο φιλόδοξη και την ενεργειακή απόδοση να τη συνδέσει σαφώς με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Γιατί αν δείτε πόσο δυναμικό υπάρχει εκεί στις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, και θα πρέπει να το συνδέσουμε με τις συζητήσεις που γίνονται για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Αλλά και στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πιο αποδοτικοί ενεργειακά και να είναι σωστή η τιμολόγηση έτσι ώστε οι νέες τεχνολογίες να οδηγήσουν σε μια νέα οικονομία που θέλουμε στην Ευρώπη και με κίνητρα έτσι, τιμών. Αυτά. Με μεγάλη χαρά να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες που θα μας κάνουν όλες τις προτάσεις και θα τους συζητήσουμε τελικά με τον Ματίας και τη Ρωμάνα Τζόρδαν, Σίσιλ να στείλουμε και ένα σαφές μήνυμα για το μέλλον, για τους κλιματικούς στόχους και ε, τους νέους στόχους για μια νέα βιομηχανική επανάσταση. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Ήταν σαφέστατες αυτές οι εξηγήσεις ε, και μας περιγράψετε το περιεχόμενο της έκθεσης και οριοθετήσατε και τη συζήτηση. Θέλουμε στα διάφορα πάνελ να καλύψουμε πολλά θέματα. Όλα αυτά που μας παρουσιάσατε και από την έκθεσή σας. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Ντόναλη, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχω στην σημερινή αυτή συζήτηση. Θα ήθελα καταρχήν να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για το σχέδιο ενεργειακής αποδοτικότητας που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα. Ταυτόχρονα σχεδόν με το σχέδιο για την οικονομία με χαμηλή χρυσή άνθρακα 2050. Άλλωστε είναι αλληλένδετα τα δύο έγγραφα. Και μάλιστα η... τα επιτεύγματα για τη χαμηλή ενέργεια του 2050 το 2020 μάλλον θα, έχουν, θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε το στόχο για το 2050 και να υλοποιήσουμε το, το στόχο της μείωσης του 20% μέχρι το 2020 και λέμε στο έγγραφο ότι αν υλοποιήσουμε του στόχους ε, για την ενεργειακή αποδοτικότητα θα καταλήξουμε σε 25% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και όχι μόνο 20%. Και μια και μιλούμε πολύ για την ενέργεια αυτό το τελευταίο καιρό και για τα συναφή θέματα, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ότι ο ασφαλέστερος ε, ε, και η ασφαλέστερη και φθηνότερη πηγή ενέργεια είναι ενέργεια που δεν χρησιμοποιούμε. Και αυτό είναι ε, απαραίτητο στοιχείο της φιλοσοφίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα και συμβάλλει και στην υλοποίηση των κλιματικών μα στόχων, αλλά και στην υλοποίηση των οικονομικών μα στόχων. Μία βιομηχανία που είναι αποδοτική και αποτελεσματική είναι ανταγωνιστική, αλλά και οι καταναλωτές έχουν όφελος ε, για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Υπάρχει εδώ και ένα οικονομικό μήνυμα πέραν του κλιματικού δηλαδή και του περιβαλλοντικού. Το σχέδιο της περασμένης εβδομάδας δίνει κάποιους προσανατολισμούς για την ενεργειακή αποδοτικότητα που υπερβαίνουν τον χρονικό ορίζοντα του 2020 και ελπίζουμε ότι δεν θα περιοριστεί εκεί και πολλές πρωτοβουλίες του σχεδίου μας θα μας βάλουν σε ένα μονοπάτι για το 2050 που θα είναι προοδευτικό, σταδιακό ε, αλλά νομίζω ότι μας δίνει τη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να τον ακολουθήσουμε ευφυώς. Έχουμε φυσικά και τα, τα σχέδια από το 2006 που συνεχίζονται. Είχαμε τις οδηγίες Σοβεζό και τις οδηγίες για τα κτίρια που ενεκρίθησαν πέρυσι. Αλλά θα κάνουμε και ένα βήμα παραπέρα. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα σημεία αυτού του σχεδίου. Θα ήθελα να πω ευθύς εξ αρχής ότι δεν υπάρχει νομικά δεσμευτικό στόχος για τη μείωση του 20% για τα κράτη-μέλη στο σχέδιο αυτό. Έχουμε όμως μία διτή προσέγγιση στο διάλογο με τα κράτη-μέλη σε δύο φάσεις. Έχουμε φυσικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να υποβάλουν ε, τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης. Θα γίνει τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο, και ω τμήμα του Εθνικού προγράμματο Μεταρρύθμισης τα κράτη-μέλη μπορούν να υποβάλουν του εθνικού του στόχου σε σχέση με του πέντε στόχου που θέτει η στρατηγική το 2020. Φυσικά έχουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη μείωση του 20%, τι ανανεώσιμε, τι κλιματικέ αλλαγέ, που είναι ε, νομικά δεσμευτικά και στα θέματα της ενεργειακής αποδοτικότητας έχουμε το στόχο του 20%. Πολλές, πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για το τι σημαίνει αυτός ο στόχος, ποιο είναι το περιεχόμενο. Στο σχέδιο προσδιορίζουμε ότι μιλάμε για πρωτογενή ενέργεια και για 368 ε, εκατομμύρια τόνους ε, μέχρι το 2050. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για δεικτικούς στόχους για τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι το 2013 θα γίνει μια αναθεώρηση, με επανεξέταση μάλλον της πρόοδου και αντίστοιχα θα προβλέψουμε ίσως και δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη-μέλη αν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νομικά δεσμευτικοί στόχοι όπως σας είπα, γιατί σκεφτήκαμε τι είναι καλύτερο, στόχους νομικά δεσμευτικούς ή μέτρα νομικά δεσμευτικά. Το σχέδιο προβλέπει νομικά δεσμευτικά μέτρα. Για αυτό θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Ότι τα μέτρα είναι νομικώ δεσμευτικά και όχι οι στόχοι. Πρόκειται για μέτρα που θα περιληφθούν στην νομοθετική πρόταση που ευελπιστούμε ότι θα καταθέσουμε τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για μέτρα που θα προβλέπουν στόχους στον δημόσιο τομέα διπλασιασμό ε, του στόχου ανακαίνηση ε, για τα κτίρια, ώστε να φτάσουμε τα 3% το χρόνο για τα δημόσια κτίρια. Επίση, ε, προσδιορίσαμε κάποια βασικά στοιχεία των κανόνων για τι κρατικέ προμήθειες και εφαρμο... της εφαρμογής γιατί οι κρατικέ προμήθειες είναι μεγάλο τμήμα τη οικονομία, ο κρατικό κλάδο, γενικώ ο δημόσιο κλάδο, και η ενεργειακή αποδοτικότητα θα πρέπει να είναι σημείο κλειδί ό,τι αφορά τι δημόσιε προμήθειε για τα αγαθά και τις υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο είναι αντικείμενο δημοσίων προμηθειών τέλος πάντων. Ο δεύτερος κλάδος δεσμευτικών μέτρων είναι η υποχρεώση εξοικονόμησης. Γιατί? Για δύο λόγους. Καταρχήν, με βάση την εμπειρία που συλλέξαμε σε πέντε κράτη-μέλη, διαπιστώσαμε ότι αυτός Δεύτερο μηχανισμός είναι αποτελεσματικός. οτι αυτος ο μηχανισμος ειναι αποτελεσματικος εχω μια ρυθμισμένη αγορά και ορατά αποτελέσματα. Το πιο σημαντικό πάντως είναι ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι κάτι που ε, καλύπτει τους πάντες. Όλοι, μπορεί να συμμετέχουν ενεργά, ιδιαίτερα οι καταναλωτές και αυτοί που μένουν στα σπίτια τους, αυτοί που εργάζονται στα γραφεία τους. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Είναι τεράστιο το φάσμα λοιπόν, γι' αυτό και είναι μεγάλη πρόκληση. Γι' αυτό και οι πάροχοι υπηρεσιών ενέργειας, επειδή έχουν τις διασυνδέσεις, το δίκτυο διανομής, έχουν την επαφή με όλο το κοινό, λοιπόν, έχουν κεντρικό ρόλο και θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά και είναι σημαντική γέφυρα ε, που μας ενώνει με τόσο πολύμορφο ακροατήριο στην Ευρώπη. Έτσι θα έχουμε τα κριτήρια και τις προδιαγραφές. Επίσης, με βάση τη συζήτηση για το σύστημα εμπορίας εκπομπών, ερχόμαστε στο νευραλικό θέμα των εκπομπών. Έχουμε φυσικά την οδηγία για τις εκπομπές, επίσης την απέτηση για την εφαρμογή της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, κάτι σχετικά καινούριο βέβαια, αλλά πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι η εφαρμογή της καλύτερης δυνατής τεχνολογίας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση οποιασδήποτε μονάδας παραγωγής ενέργειας θα πρέπει να είναι σημαντική όχι μόνο όταν ε, κατασκευάζεται ένα νέο εργοστάσιο, αλλά και για τα ανανεώσιμα, γιατί υπάρχει πενταετής κύκλος και εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιείται καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία. Βέβαια είναι κάπως προβληματικός αυτός ο κλάδος και ο τομέας μάλλον και εκεί που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτή η απέτηση για τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες μπορεί να παρακαμφθεί από τις ε, βιομηχανίες που εμπίπτουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Γιατί το σύστημα αυτό που περισσότερο καλύπτει τις εκπομπές άνθρακα δεν είναι το καλύτερο εργαλείο για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν είναι ίδιοι στόχοι λοιπόν, παρόλο που είναι ελλοσυμπληρούμενοι, αλλά η ιδέα της εξαίρεσης ε, Όλε τι βιομηχανίε που εμπίπτουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών από τι απαιτήσει ενεργειακή αποδοτικότητα δεν έχει νόημα κατά τη γνώμη μα και αυτό το αναφέρουμε στην πρόταση. Ένα άλλο αλληλεύθερο θέμα είναι και το θέμα τη θέρμανσης. Θέρμανση για τα κτίρια. Το κτίριο που βρισκόμαστε, αυτά που βλέπουμε στο παρά, από το παράθυρο, τα σπίτια μα, που είναι το 40% της ενέργειας που καταναλώνουμε στην Ευρώπη. Η ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των κτίριων. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη δαπάνη ενέργειας που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κεντρικό τομέα που θα πρέπει να καλύψουμε με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ο πρώτος και πιο σημαντικός και ο πιο σημαντικός μηχανισμός που έχουμε είναι να εξασφαλίσουμε ε, ότι το περίβλημα ενό κτηρίου είναι ασφαλέ και αποτελεσματικό. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο βέβαια για τα νέα κτίρια, γιατί ξεκινάμε από τα θεμέλια και το κόστος μπορεί να είναι συμπληρωματικό, αλλά δεν είναι τόσο, τόσο μεγάλο όσο στην ανακαίνιση των ε, κτηρίων που ήδη ε, υπάρχουν. Βλέπουμε απέναντι, από το, απέναντι μας σπίτια που μπορεί να είναι και 80 και 100 ετών. Το θέμα είναι πώς θα εξασφαλίσουμε και σε αυτά τα παλιά κτίρια, σε αυτά τα παλιά διαμερίσματα που, λέμε, που βλέπουμε, να εξασφαλίσουμε ε, και το περίβλημά τους να είναι ασφαλές. Βέβαια αυτό είναι πολύ πιο δαπανηρό, αλλά απαραίτητο για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Και πώς θα αποδεσμεύσουμε κάποια κονδύλια, πώς θα βρούμε κονδύλια για τη χρηματοδότηση. Εδώ μιλούμε για τάξη μεγέθους ε, τεράστια για κονδύλια. Ξεπερνάει οποιοδήποτε στόχο δημοσιονομικών προοπτικών. Σίγουρα δεν μπορούμε από τις δημοσιονομικές προοπτικές να βρούμε αυτά τα κονδύλια. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να ε, έχουμε κάποιες δράσεις υποστήριξης μέσω χρήσης ε, των διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας ε, προς την ενεργειακή αποδοτικότητα και με αποκεντρωμένο τρόπο να χρηματοδοτήσουμε κυρίως αυτή την ε, ανακαίνιση των κτίριων. Ένας άλλος τομέας στο δημόσιο επίσης αφορά τη χρηματοδότηση του κόστους για την ανακαίνιση των κτίριων. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια προβλήματα στους κρατικούς προϋπολογισμούς και λιτότητα. Θέλουμε προβολή, νομιμοποίηση και υποστήριξη των συμβάσεων για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Οπότε ο εργολάβος να χρηματοδοτεί με αποτελεσματικό τρόπο την επένδυση και ε, να μπορεί να αποσβένει αυτή την ε, ε, επένδυσή του σε 10-20 χρόνια. Γνωρίζουμε ότι σε πολλές χώρες μέλη έχουμε δυστυχώς ανυπέρβλητα εμπόδια. Νομοθετική διαδικασία καταρχήν που χρησιμοποιείται για τις δημόσιες προμήθειες που δεν επιτρέπει τέτοιες δεκαετίες, 20 ετής συμβάσεις. Αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά και κανόνες για τα λαγιστικά που λένε συνήθως 100 μονάδες σε πέρυσι, 80 φέτος, αναφέρονται 80 στον προϋπολογισμό. Είναι δύσκολο να υπολογιστεί η απόσβεση. Θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση και των εθνικών λογιστικών κανόνων, λοιπόν, για να επιτρέπονται τέτοιες ίδιους μακροπρόθεσμες ε, συμβάσεις. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, επαγρύπνηση, συνειδητοποίηση γιατί χρειαζόμαστε χρηματοδότηση των επενδύσεων από τις κεφαλαίες αγορές. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που χρησιμοποίησαν ένα κονδύλιο των, του πακέτου ανάπτυξης για το Ειδικό Ταμείο Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Και μάλιστα ελπίζουμε ότι μέσα σε ένα μήνα να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το χρηματοδοτικό μέσο στο Λουξεμβούργο. Το υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το έχει περικοδοτήσει με κάποια κονδύλια. Και μάλιστα προσκαλέσαμε και άλλες δύο τράπεζες να συμμετέχουν σε αυτό το ταμείο και ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε τη μόχλευση ώστε να έχουμε ένα ταμείο 500, 600 εκατομμυρίων που θα υποστηρίζει ευρώ, που θα υποστηρίζει αυτά τα μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και θα βοηθήσουμε και τις τοπικές αρχές στις προσπάθειές τους ε, να υλοποιήσουν τέτοιους στόχους. Το σχέδιο περιλαμβάνει και άλλα θέματα βέβαια. Προσπάθησα να είμαι πιο συνοπτική. Τώρα Προσπαθούμε να συνδυάσουμε το πακέτο αυτό με τους κλιματικούς και τους οικονομικούς μας στόχους. Και φυσικά με πρωτοχικό στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ εύγλωτα όλα αυτά. Μας αναφέρατε διάφορες προσεγγίσεις που μας είναι πολύ χρήσιμες για τη δουλειά μας, τις κλιματολογικές αλλαγές σε σύνδεση με τα οικονομικά. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πριν αρχίσει η συζήτηση εδώ ότι αυτές τις μέρες συζητάμε και ένα θέμα σχετιζόμενο με αυτό τις προτεραιότητες στις ενεργειακές υποδομές. Γιατί με υποδομές δεν εννοούμε μόνο για τις μεταφορές των διαφόρων τρόπων ενεργείας αλλά και την, τα δίκτυα διανομής των Συνήθως μιλάμε για τα λεγόμενα έξυπνα δίκτυα ή smart grids και είναι θέμα και αυτό που πρέπει να το θίξουμε γιατί είναι θέμα εξοικονόμησης και καλύτερης χρήσης αλλά και πρέπει να δούμε και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να ανανεωθεί, θα μπορούσαν να ανανεωθούν τα υπάρχοντα δίκτυα διανομής. Υπάρχει το θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ο αναποτελεσματικός τρόπος κατανάλωσης ενεργείας. Για όλα αυτά χρειαζόμαστε τα smart grids, τα έξυπνα δίκτυα. Η Κομισιόν το ξέρει το πρόβλημα και εμείς πρέπει να το ξέρουμε όμως. Σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις βέβαια για να λυθεί το πρόβλημα αυτό για το μέλλον και όποτε μιλάμε για ενεργειακή αποτελεσματικότητα ή εξοικονομήσεις δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ένα σχόλιο αυτό ήταν απλώς για να προσθέσω σε αυτά που είπε η ομιλήτρια και έχετε το λόγο τώρα όσοι θέλετε να μιλήσετε. Η Λίνα Εκ από τους συναντέλφους έχει ζητήσει το λόγο και ο Μπένσον βέβαια. Ορίστε Λίνα πρώτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αντώνηλη. Εννοώ ότι ευχαριστώ και τους συναδέλφους βέβαια, αλλά με τους συναδέλφους. Χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί η Κομισιόν τελικά καταλαβαίνει αντιλαμβάνεται τις προτάσεις αυτές όπως και εμείς τελικά. Χρειάστηκε μεγάλος αγώνας για να κρατηθούν ορισμένα ποσά για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Να δοθούν λίγα και για τους πολίτες. Διότι φαίνεται ότι τελικά βρίσκονται τα χρήματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότατα. Επειδή τους τελευταίους μήνες βρέθηκαν χρήματα, τα βάλαμε όλα σε αυτό το ταμείο. Και όταν θα λυθεί θα ανοίξουμε μια σαμπάνια. Για την ενεργειακή αποδοτικότητα έχω συναντηθεί με εκπροσώπους της Euroelectric οι οποίοι ανησυχούν ότι μήπως ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεστε το θέμα κατακαιρματίσει την αγορά. Δεν είναι κατά του 30% αλλά θα ήθελαν μια πιο προβλέψιμη καμπύλη να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στην μέθοδο εργασίας σας λοιπόν πώς φροντίζετε να μην κατακαιρματιστεί η αγορά γιατί υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα σε κάθε χώρα μέλος δεν υπάρχει ενιαία εσωτερική αγορά ενεργείας που αποφασίσαμε να δημιουργηθεί. Γιατί εδώ δεν έχουμε καθορίσει ούτε καν ευρωπαϊκούς στόχους. Πόσο μάλλον ανατομέα και χώρα. και ίσως αυτό να μην προσθέτει καθόλου ανταγωνιστικότητα. Δεύτερο ερώτημα. Σε μερικές χώρες η ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση και την ψήξη έχει αγνοηθεί. Τρίτον, για τις ατομικές καταμετρήσεις. Έχουμε πει να υπάρχουν μετρητές, αλλά χωρίς να αναφέρουμε ποια θα είναι η τιμή τους. Ο καταναλωτής και η καταναλώτρια θα έχει λέει τη δυνατότητα να επιλέγει το δίκτυο, να γνωρίζει πόσο καταναλώνει αλλά δεν δίνουν όλες οι εταιρείες σαν την ΕΝΕΛ πλήρεις πληροφορίες για τις τιμές τους και τις ταρίφες τους. Γιατί όταν ξέρουμε σε ποια ωράρια είναι η φτηνότερη τιμή, το εκμεταλλεύεται αυτό ο καταναλωτής και η καταναλώτρια. Όταν θα εγκατασταθούν οι μετρητές θα φανεί αυτό καθαρότερα. Γιατί θα ωφεληθεί και το δίκτυο και ο καταναλωτής και θα υπάρξει μεγαλύτερη αποδοτικότης. Εσείς εκεί κάτω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε λέει ο μιλητής. Είναι μεγάλη χαρά η παρουσία μου εδώ απόψε. Και μου άρεσαν επίσης και τα σχόλιά σας για την ενεργειακή αποδοτικότητα που ξεπερνούν ακόμη και τους στόχους που είχαμε θέσει για το 2020 τα 5 τα 500 με 600 εκατομμύρια που προβλέπονται εδώ ε, είναι ίσως ψηλό ποσό γιατί δεν είμαστε βέβαιοι πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν. Πω, ρωτώ, πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα αυτά κύρια Κομισιόν. Έχετε καμία περαιτέρω εξήγηση. Καμία. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα χρησιμοποιήσετε τα χρήματα. Ο Μπάσεκ Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη Μαρή για την εισαγωγή στην ενεργειακή απόδοση, οικονόμηση ενέργειας και ε, που τονίσατε και τη σημασία. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μας δείχνει η έρευνα ότι ε, ε, πρέπει να φτάσουμε στους στόχους μας, αλλά έτσι όπως το πάμε, αν δείτε τα στοιχεία, θα είμαστε στο 9% μέχρι το 2020, αντί το 20%. Το λένε σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση. Παλιά το λέγανε πρόγραμμα δράσης. Η δράση έχει φύγει, έχει μείνει το πρόγραμμα μόνο. Πολύ εύγλωτο και αυτό. Τα επόμενα χρόνια, δεν μιλώ τώρα για τη δημόσια συμβάση και τα κρατικά κτίρια, διότι εντάξει ωραία είναι όλα αυτά, αλλά για να είμαστε ειλικρινεί, τα περισσότερα κτίρια που καταναλώνουν ενέργεια δεν είναι δημόσια. Εντάξει, να αρχίσετε από τα κρατικά, αλλά υπάρχουν και άλλα και τι θα προτείνετε για να βεβαιωθείτε ότι ο στόχος του 20% θα φτάσει πιο κοντά μας από το 9% που λέμε. Γιατί αν περιμένουμε μέχρι το 2013 και μετά θα κάνετε την ανάλυση αν και κατά πόσο προχωρούμε και μπράβο και αν συνεχίσουμε όπως τώρα μπορεί το 2013 να έρθείτε να ε, συμπεραίνετε ότι χρειάζονται πιο επιθετικές πολιτικές όλα αυτά ωραία και μετά θα μας πείτε ότι για να εγκριθούν πρέπει να είναι το 2014. Βλέπε ευρωεκλογέ, νέο κοινοβούλιο, νέα κομισιόν και πριν ε, ε, έρθει η νέα νομοθεσία, χαιρετίσματα. Πάμε στο 15 και στο 16. Και ακόμα παραμένουμε στο 20% μέχρι το 2020 για τόσο σημαντικά στοιχεία που είναι η κλιματική πολιτική. Δεν μπορώ να καταλάβω τι περιμένουμε μέχρι το 2013, γιατί δεν τα κάνουμε από τώρα. Γιατί δεν αναβάλουμε τις μελλοντικέ μας πολιτικές μέχρι το 2016, γιατί ξέρουμε ότι σίγουρα τότε δεν πρόκειται να φτάσουμε στο 2020 το 20%. Είναι θεωρητικό στόχος και μόνο. Ευχαριστώ. Η Αντίτια Τσόκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επιτροπή μας που διοργανώνει αυτή τη ενδιαφέρουσα συζήτηση και ε, όλοι οι βουλευτές που ενδιαφέρονται για την ενέργεια είναι παρόντες. Οι υπόλοιποι έχουν ήδη πάει για Σαββατοκύριακο, από ό,τι φαίνεται. Η κυρία Ντόνελη είπε ότι η πιο φτηνή ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνουμε. Μα χρειάζεται και κάποια εγκατάσταση για την εξοικονόμηση και για την απόσβεση της εγκατάστασης αυτής της επένδυσης είναι μία δεκαετία. Και παραπάνω. Δηλαδή μέχρι να φτάσουμε να εξοικονομούμε ενέργεια έχουμε κάνει μια επένδυση που έχει ένα κόστος και χρειάζεται δεκαετία για να αποσβεστεί. Εντάξει, από εκεί και πέρα ε, φυσικά η πιο φτηνή ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνουμε, αλλά το δίκτυο τι θα το κάνει. Να ξανάρθω εγώ στο αγαπημένο μου θέμα τι γίνεται με την επαγγελματική κατάρτιση για ε, κλάδους που δεν παράγουν διοξίδιο του άνθρακα. Ε, κάθε μικρομεσαία επιχείρηση πρέπει να έχει αναλογιστεί για να δει πώς μπορεί να εξοικονομεί χρήματα και να διαχειρίζεται την οικονομία της. Ωραία. Έχουν ταυτόχρονα όμως και έναν ειδικό για την ενέργεια, για να τους λέει πώς θα εξοικονομούν ενέργεια εκτός από λεφτά. Απάντηση όχι. Και όσο δεν υπάρχουν τέτοιοι ειδικοί, δεν ξέρουν και εταιρείε τι να κάνουν. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να απαντηθεί αυτό στις δεξιότητες, στα προσόντα, στην επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρώπη. Κάποιο άλλο το είπα ε, επίσης. Είναι πολύ μεγάλη αναντιστοιχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που λέμε και αυτό που κάνουμε. Αν κάποιος δεν μιλήσει για ενεργειακή απόδοση, σε κάποιες χώρες της Ένωση θα χάσει τι εκλογές. Σε άλλες μόλις το ξεστομίσει θα χάσει επίσης τι εκλογές. θα πρέπει να αντιστοιχούν ε, τα έργα μας με τα λόγια μα. Σε πολλές χώρες υπολείπονται αυτοί και δυστυχώ και δικιά μου ανήκει αυτές. Τώρα βέβαια μετά όσο συμβαίνει στη Βόρεια Αφρική και στην Ιαπωνία δεν το συζητάμε αλλά αλλάζουν τα δεδομένα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Στις 3 Μαρτίου ε, ιδρύσαμε και άρχισε να λειτουργεί ένα νέο οργανισμό. Το ΕΣΑΡ, τι, μπορεί να κάνει αυτό, πώς θα λειτουργεί και τι θα προσφέρει. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ. Πολλές συζητήσεις έγιναν για την εξοικονόμηση ενέργειας, για την περιβαλλοντική πολιτική, για την πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό που είναι ενδιαφέρον στη σημερινή δημόσια κρόση είναι ότι προσπαθούμε να συνδυάσουμε το κλίμα, την ενεργειακή πολιτική και τη βιομηχανική μας πολιτική. Έχω μια ερώτηση και προς την Επιτροπή, αλλά ελπίζω να το ακούσω και από τους ε, επόμενους εμπειρογνώμονες. Τα αποτελέσματα των πολιτικών μας στη βιομηχανία ποια είναι. Γιατί μας πλησιάζουν λόμπι από διάφορες βιομηχανίες που διαμαρτύρονται για τα ολέθρια αποτελέσματα της πολιτικής μας στη βιομηχανία. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, οι μελέτες που να μας ενημερώνουν για τον αντίκτυπο που έχει η πολιτική αυτή στη βιομηχανία και πώς οι επιχειρήσεις αυτές θα υποφέρουν κατά κάποιο τρόπο λόγω της αναδιοργάνωσης, ανασυγκρότησης που υποχρεούνται να υποστούν η πολιτική μας αυτή θα έχει τόσο αρνητικές συνέπειες οικονομικές που θα τους υποχρεώσει να εγκαταλείψουν την Ευρώπη. Γιατί είπε και η Λένα ότι το κεφάλαιο δεν επιλέγει την Ευρώπη για τις επενδύσεις του, προτιμάει να πάει σε άλλες υπήρους για να επενδύσει. Μήπως και αυτό οφείλεται στην ε, ενεργειακή και την κλιματική μας πολιτική ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι γι' αυτό. Σίγουρα στην Ευρώπη έχουμε ψηλότερους μισθούς από ό,τι στην Κίνα, για παράδειγμα. Και αυτό είναι αντικίνητρο για τις επιχειρήσεις. Αλλά σε ποιο βαθμό και η κλιματική μας πολιτική και η ενεργειακή μας πολιτική συντελούν στην ε, έξοδο των επιχειρήσεων. Ίσως ε, καλό θα ήταν να βολιδοσκοπήσουμε και τους ε, κύριους εταίρους μας με μεγάλες βιομηχανίες για να μας εξηγήσουν γιατί φεύγουν από την Ευρώπη. Γιατί οι χώρες που έχουν αλλοδαπό κεφάλαιο θα πρέπει να δούμε πώς το καταφέρνουν. Βέβαια, πολλές φορές αυτό οφείλεται στο άνοιγμα των αγορών και στην ελεύθερη πολιτική που έχουν. Ο Καρλ Χάιν Φλόρεντς. Ε, finde das sehr gut, dass Sie heute äh, Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται αυτή η ακρόαση σήμερα και έχουμε και εμπειρογνώμονες καλέσει. Θέλω να υποστηρίξω και το συνάδελφο Eckhout. Ε, βέβαια μπορεί να είμαστε από διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις, αλλά... Ε, Βλέπουμε αυτές τις εβδομάδες τι ζούμε, ε, όλη αυτή τη δυστυχία και τα δεινά και για μένα δεν είναι άσπρο μαύρο αυτά τα θέματα. Να ακριβίνουμε την ενέργεια για να παράγουμε λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα και έτσι αποδυναμώνουμε τις αγορές. Όχι, πρέπει να το δούμε αλλιώς. Να έχουμε επίγνωση ότι μπαίνουμε τώρα σε μια νέα εποχή ενεργειακής πολιτικής. Και αυτό είναι ευκαιρία, δεν είναι τιμωρία. Εγώ μένω σε μια χώρα όπου ένα μόσπονδο κρατήδιο ε, έχει αρχίσει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα αιωλικού πάρκου και παράγουν όχι για τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία δεν τη θέλουν αυτή την ενέργεια, αλλά εξάγουμε προς την Κίνα, πάρα πολύ στην Κίνα. Ε, γίνονται πολλές προσπάθειες, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, υπάρχει αυτή η αποσύνδεση των θεμάτων και να βγούμε λίγο με ελπίδα προς το μέρον, όχι όλα αυτά τα καταθλιπτικά που ακούμε και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτούς τους τομείς. Νομίζω ότι η Γερμανία έχει κάνει κάποιες καλές προσπάθειες, καλή αρχή βέβαια και σφάλματα δεν χωράει, καμία αμφιβολία. Αλλά ε, είναι γεγονός το εξή. Επί σειρά ετών ε, στα ομόσπονδα κρατήδια, στους προϋπολογισμούς είχαμε χρήματα τα οποία δεν απορροφούσαμε για ανανεώσιμα πράγματα. Για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι τρέχει. Ότι η σωστή και φρόνιμη διαχείριση των πρώτων υλών ε, είναι κάτι που αφορά και τα παιδιά μας. Εγώ ξέρετε δεν είμαι γενικά συναισθηματικός άνθρωπος, αλλά ε, αν κοιτάξετε τα σπίτια στις Βρυξέλλες, θα πέσετε κάτω από την κατάσταση ε, των κατοικίων. Παρόλο που αγαπάω πάρα πολύ τις Βρυξέλλες, δεν φταίνουν τα παράθυρα, φταίνουν οι διοκτήτες που δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Και θα παρακαλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε τέτοια ζητήματα να ενεργοποιείται για συνειδητοποίηση, για εκπαίδευση, για μόρφωση και ταυτόχρονα να τραβήξω και λίγο φρένο γιατί η αγαπητή μου συνάδελφος ε, από τους σοσιαλιστές θέλει να δώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τώρα και ένα αρμόδιο για θέματα ενέργειας. Ε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ και καιρό έχουμε θέμα οικολογικού λογιστικού ελέγχου, αυτό που λέμε το eco audit. Και ξέρει κανείς πόσα ε, κιλοβάτ ώρες ε, ρεύμα χρειάζεται για να φτιάξει ένα τόνο ατσάλι. Αυτά θα πρέπει να είναι ενιαία και όχι από ε, πάνω εμείς να επιβάλλουμε στις εταιρείες να προσλαμβάνουν έναν ειδικό, έναν αρμόδιο για την ενέργεια. Πού θα τα βρουν τα λεφτά εταιρείες. Και η χρηματική υποστήριξη, η κινητροδότηση οικονομική για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Τις τελευταίες ε, εβδομάδες, τους τελευταίους δύο μήνες, ε, βλέπουμε να είναι της μόδας αυτό το θέμα της εξοικονόμησης συνέργειας. Ε, πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα, εγώ δεν το αφισβητώ, αλλά δεν μπορεί κάποιοι παλαβοί υπάλληλοι στις Βρυξέλλες να καταστρέφουν τους γερμανικούς νόμους, γιατί εμείς καλέσαμε τους γερμανούς πολίτες, τους ενθαρρύναμε να εξοικονομούν ενέργεια να περάσουν στι ανανεώσιμε και επειδή κάποιοι άλλοι δεν το θέλουν, παρόλο που έχουν περισσότερο ήλιο από εμά, δεν θα καταστρέψουμε την πολιτική μα. Και αυτό δεν το έφερε η δική μου κυβέρνηση. Το έφερε μια κυβέρνηση σοσιαλιστών και πρασίνων που δεν είναι και αγαπημένη μου. Αλλά δεν θα πρέπει να καταστρέφουμε τέτοιε προσπάθειε, να τι διορθώνουμε. Ευχαριστώ, Καρλ Χάιντ. Ο κύριο Γκέμπελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί, κυρίε και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτιαξε αυτή την περίφημη στρατηγική για το 2020. Τη χαρακτηρίσαμε φιλόδοξη και είχαμε και το φιλόδοξο στόχο να συμπαρασύρουμε και το υπόλοιπο κόσμο. Είδαμε το αποτέλεσμα στην Κοπεχάγη, πλήρες ναυάγιο. Και το υποτιθέμενο αποτέλεσμα το διαπραγματεύτηκαν άλλοι. Και η Μέρκελ, ο Σαρκοζή και ο Μπαρόσο ήταν έξω από την αίθουσα. Τα έκαναν οι, Κινέζοι, οι Νοτιοαφρικανοί, οι Βραζιλιάνοι, οι Αμερικανοί κτλ. Συνεχίστηκε η προσπάθεια στην Κανκούν με το αποτέλεσμα που γνωρίζουμε, δηλαδή μηδαμινό. Δέσμευση, εντάξει, ότι στόχος είναι το 20% ή το 2% μάλλον δύο βαθμοί εννοεί ο μιλητή. λες και είναι θερμοστάτη στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα και το κατεβάζει δύο βαθμούς. Οι συνολικέ εκπομπές ρήπων λοιπόν, των 27 κρατών μελών είναι γύρω στο 11% των παγκοσμίων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. 18 είναι οι χώρες στον κόσμο αυτό που εκπέμπουν 80% των συνολικών ρήπων. Μεταξύ αυτών των 18 είναι μία ε, ε, ευρωπαϊκή χώρα, η Γερμανία, η μεγαλύτερη και πιο βιομηχανική. Εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι με μονομερείς δράσεις η Ευρώπη θα μπορέσει να συμπαρασύρει και τα άλλα κράτη. Εμείς ε, θέλουμε δεσμευτική συμφωνία, διεθνή συμφωνία. Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να την αποκτήσουμε. Αλλά για τον εξή απλούστατο λόγο, ότι η Κίνα σιγά μην κάτσει να την κλείσουμε σε ένα τέτοιο τέλμα. Και αν δεν το κάνει η Κίνα δεν θα το, την ακολουθήσουν ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι υπόλοιποι. Ε, η Ρωσία, η Ινδία, η Βραζιλία κλπ. Αυτό είναι πραγματικότητα και νομίζω αναφυσβήτητη. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν προσπάθειες και οι χώρες αυτές. Η Κίνα μόλις υιοθέτησε ένα πενταετές ε, ε, πρόγραμμα που ε, χαιρέτησε ε, η κυρία Χίλντεγκαρτ τεχτέ, αν ε, διάβασα σωστά τον τύπο. Κάνει πολλέ προσπάθειες η Κίνα, φιλότιμες, για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, αποδοτικότητα, ό,τι θέλετε να εξοικονομήσει. Όλα αυτά τα πολύ αξιέπαινα που θέλουμε κι εμεί να κάνουμε. Και άλλες χώρες ακολουθούν. Η Κίνα μάλιστα από πέρσι έγινε ο πρώτο παγκόσμιο εξαγωγέ ανεμογεννητριών και ολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών. Αυτό τι αποδεικνύει, ότι η τεχνολογία, η κινέζικη τεχνολογία εγώ, είναι μάλλον ε, ανώτερη ή εν πάση περιπτώσει φθηνότερη από την ευρωπαϊκή τεχνολογία που θέλουμε να κάνουμε εμείς λέει την πράσινη επανάσταση. Αλλά οι στόχοι ε, των άλλων και των Αμερικανών και των Κινέζων είναι πενταετίας. Εμείς έχουμε ένα ορίζοντα μέχρι το 2050 και αναρωτιόμαστε αν θα είμαστε στο 90% των ανανεώσιμων ή στο 100%. Πολύ σοβαρά όλα αυτά. Αφήστε δε που το 2050 δεν θα υπάρχει κανείς από εμά όλους εδώ τους σημερινούς ε, ε, νομοθέτες που παίρνουν τις αποφάσεις δεν θα είναι κανείς για να ελέγξει αν όλα αυτά έγιναν πραγματικότητα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ε, για τα γεγονότα στην Ιαπωνία, τα οποία δεν συζητούμε κατά τα άλλα σήμερα, ότι θα μειώσουν τη παραγωγή πυρηνική ενέργεια τουλάχιστον στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, στην Κίνα και αλλού ενδεχομένω όχι, αλλά στην Ευρώπη οπωσδήποτε. Αυτό τι σημαίνει. Αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρώπη, που κάπω πρέπει να τις αντισταθμίσουμε, δεν ξέρω πώς. Βεβαίως να επενδύσουμε σε ανανεώσιμε. αλλά όταν μιλάμε για ενεργειακή απόδοση, τι σημαίνει αυτό. Η ηλιακή ενέργεια είναι αποδοτική, είναι ενέργεια που μας επιτρέπει να κάνουμε οικονομίες, τουλάχιστον όχι στη Γερμανία και σε χώρες όπως τη δική μου, όπου η ηλιοφάνεια είναι 800 ώρες περίπου το χρόνο. Ενώ στην Ισπανία είναι 2.000 ώρες το χρόνο και στη Βόρεια Αφρική 2.500 ώρες. Ας είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές. Συμφωνώ να επενδύσουμε στην ενεργειακή απόδοση και όλα αυτά τα ωραία που λέτε ε, ε ως απαραίτητα. Την ανακαίνιση των κτηρίων. Ε, το κάνουμε όμως. Αντί να επενδύουμε σε διάφορα gadgets. Και θα σταματήσω εδώ. Αντί να έχουμε όλο και περισσότερους θεωρητικούς στόχους, Ας επικεντρωθούμε, ας συγκεντρωθούμε σε αυτά που είναι σήμερα εφικτά και την επόμενη πενταετία. You, uh, Ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε τρία πάνελ στη Δημοσία κρόση και αυτό είναι το εισαγωγικό πάνελ. Ας μην επεκταθούμε υπερβολικά λοιπόν. Το λόγο θα δώσω στην κυρία Ντόναλη, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο εισαγωγικό πάνελ και να περάσουμε στα πάνελ των εμπειρογνωμόνων. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας. Ελπίζω να μην ξεχάσω καμία, αλλά θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω. Τέθηκαν ερωτήσεις για το πακέτο ανάκαμψης και τι γίνεται με τα κονδύλια που είχε προβλέψει. Τώρα οριστικοποιούμε πολλά γραφειοκρατικά με την ΕΤΕ και με τις αρχές του Λουξεμβούργου, προκειμένου να ιδρύσουμε το επενδυτικό ταμείο και να μεταφερθούν τα κονδύλια από την ΕΤΕ στο επενδυτικό ταμείο. Και ελπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και οι επενδυτικές κατευθυντήρες γραμμές προβλέπουν επικέντρωση στην ενεργειακή απόδοση. Καλύτερη ε, ανακαίνιση και αποτελεσματικότερα κτίρια και υποστήριξη των τοπικών αρχών. Θέλουμε να στηρίξουμε τις τοπικές αρχές και τις αρχές των πόλεων και τα αστικά κέντρα για να επενδύσουν σε αυτό το θέμα της ενεργειακής απόδοσης. Αν κάποιος θέλει περισσότερες λεπτομέρειες, πολύ ευχαρίστως, γιατί πραγματικά αυτό το ζήτημα είναι φλέγον. Ως προς τη βιομηχανία, θα ήθελα να πω ότι η βιομηχανία στην Ευρώπη, αν ρίξετε μια ματιά στην ανάλυση και τις μελέτες που κάναμε, είχε τις καλύτερες επιδόσεις ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Γιατί εξετάζουμε τρει τομείς συνήθω. Αλλά η βιομηχανία από τους τρει είναι αυτή που έχει την καλύτερη εξοικονόμηση, τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτή την εξοικονόμηση ενέργεια και δεν μα εκπλήσει αυτό γιατί είναι λογικό, φυσιολογικό να κάνει οικονομίε η βιομηχανία. Αλλά η βιομηχανία απαρτίζεται από τρει μεγάλες ομάδες. Έχουμε τη βιομηχανία που παράγει ενέργεια και καλύπτεται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Έχουμε βιομηχανία με μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά όχι αρκετά μεγάλες ό,τι αφορά τη χρήση ενέργειας. Δηλαδή έχουν ενεργειακό κόστος, αλλά δεν είναι το βασικό τους κόστος. Και έχουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε όσους παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και εμπίπτουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, ήδη είπα ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών από μόνο του δεν είναι το πιο εκλεπτισμένο εργαλείο για την ενεργειακή απόδοση και θα πρέπει να το ενισχύσουμε με κάποιο τρόπο. Για τις μεγάλες εταιρείε που έχουν ενεργειακό κόστος αλλά δεν είναι το μείζον κόστος τους, το σχέδιο προβλέπει υποχρεωτικούς ενεργειακούς ελέγχους γιατί ε, θα πρέπει να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι και είπαμε να, γίνει, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος το κόστος το ενεργειακό. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν προτείνουμε τέτοιους ελέγχους γιατί πραγματικά αυτό θα είναι αβάσταχτο άχθος για αυτές, αλλά προτείνουμε καλύτερη ενημέρωση και συνεργαζόμαστε με τη σωματεία τους και τις οργανώσεις για να γίνουν εδώ είδος συγκριτικής των τύπων βιομηχανικών παραγωγών, με τους αρτοποιούς για παράδειγμα. Ε, ενημέρωση ως προς την ενεργειακή απόδοση των φούρνων. Ένα είδος benchmark συγκριτικής αξιολόγηση, ένα πλούστατο εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν στοιχίζει τίποτα και τους ενδιαφέρει άμεσα. Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε είναι οι έξυπνοι μετρητέ. Πολύ σημαντικό ζήτημα, όχι μόνο για τους καταναλωτές, κυρίως βέβαια για τους καταναλωτές, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι ευφύες μετρητέ είναι το καλύτερο εργαλείο που μπορεί να έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αλλά χρειάζεται σωστή ενημέρωση με ευανάγνωστο, εύληπτο τρόπο και δεν χάζει οι επιχειρηματίες, αυτοί που έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σωστή ενημέρωση μπορούν να ανταποκριθούν. Και με τους ευφύς μετρητές θέλουμε να εξασφαλίσουμε πρώτα-πρώτα τη λειτουργικότητά τους. Δεν λέμε θα πάρετε ένα ή ένα ένα κόκκινο, ένα μπλε μετρητή, αλλά να πούμε ότι ο μετρητή θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτέ τι πληροφορίε. Θα πρέπει να είναι προσιτό με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να κάνει επιλογέ ανάλογα με το στόχο. Λειτουργικότητα λοιπόν και διάφορες λειτουργίες που προσδιορίζουν τη χρήση του εφιούς μετρητή. Και οι υπάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών θα μπορούν να υποστηρίξουν και το, την παροχή των εφιών μετρητών, που επαναλαμβάνω θα είναι πολύ χρήσιμη και για τους καταναλωτές και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προετοιμάζουμε τώρα κάποιες νομοθετικές προτάσεις. Και μάλιστα ο συνάδελφος εδώ θα έπρεπε να είναι στο γραφείο του και να οριστικοποιεί το κείμενο, γιατί το ετοιμάζουμε και θα το υποβάλουμε τις επόμενες εβδομάδες. Και ε, η αισιοδοξία μας υπαγορεύει ότι είναι προτεραιότητα ως νομοθετική πράξη και <laughs> ότι θα περάσει από το Συμβούλιο και θα και στην πρώτη ανάγνωση. Αυτό μας λέει μια αισιόδοξη προοπτική. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάντως είναι να αναλάβουμε ανυπερθέτως δράση με νομοθετικά μέτρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το 2013 ή ακόμη πιο πέρα, πιο αργά, για να θεσπίσουμε νομοθετικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά τις ε, πολυμερείς και μονομερείς συμφωνίες, οι διμερείς συμφωνίες. Συμφωνώ με αυτό που είπατε για την Κίνα. Είχαμε συναντήσει με Κινέζους εκπροσώπους και μας εξήγησαν το περιεχόμενο του πενταετούς του πλαισίου. Το πιο ενδιαφέρον είναι τα κίνητρα που δίνονται στην Κίνα για την ενεργειακή απόδοση, ιδιαίτερα στη βιομηχανία, που πραγματικά έχει οικονομικό προσανατολισμό. Και η θέση τους είναι απλή. Γνωρίζουν ότι έχουν ένα ανταγωνιστικό ε, πλεονέκτημα σήμερα σε ό,τι αφορά τους μισθούς Βέβαια, γνωρίζουν ότι όσο περνάει ο χρόνο θα αποδυναμώνεται αυτό το πλεονέκτημα, γι' αυτό αναζητούν άλλους τρόπους. Και μια και που η παιδίση είναι καινούργια ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας και τις υποδομές, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αιχμή της ε, απόδοσης και θεωρούν ότι η ενεργειακή απόδοση θα τους αυξήσει το, ενεργεια... το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Και νομίζω ότι πολλά μπορούμε να διδαχθούμε από την κινέζικη αυτή ε, προσέγγιση. Γιατί πραγματικά το σχέδιο ενεργειακής απόδοσης θα μας ε, βοηθήσει να υλοποιήσουμε όχι μόνο τους κλιματικούς μας στόχους, αλλά και τους οικονομικούς μας στόχους. Αυτά και ελπίζω να απάντησα. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε τώρα με το πρώτο πάνελ. Θα αλλάξει η Προεδρία, θα δώσω τη σκητάλη στο Ματίας. Σας ευχαριστώ. Und ich muss als erstes noch Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω, ε, οφείλω να καλωσορίσω, αλλά θέλω και να καλωσορίσω ε, μια ομάδα επισκεπτών, ε, Φαγέτ College από τη Βρέμη, είναι νέοι ε, ε Αμερικανοί, ε, ως και νέες φοιτητές και φοιτήτριες και χαίρομαι ε, που ε, συμμετέχουν σήμερα εδώ στη ε, συνεδρίασή μας και στην ακρόαση μας. Καλώς ορίσατε και παρακαλώ τους εμπειρογνώμονες να έρθουν στο πάνελ. Λοιπόν, αρχίζουμε. Πρώτος εμπειρογνώμων είναι ο κύριος Ματίας Ντίνχαρτ από την εταιρεία Rhein Energy και θα μας μιλήσει για την εξοικονόμηση ενέργειας και ε, το δυναμικό των λεγόμενων πρασίνων θέσεων απασχόλησης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε στα αγγλικά. Κυρίες και κύριοι, Καλημέρα σας. Λέγομαι Ματία Δίνερτ, είμαι από τη Rhein Energy που είναι μια μεσαία επιχείρηση ενέργειας στη Γερμανία. Δεν είναι γίγας αλλά ούτε και νάνος από εταιρείε. Δεν θα σας δείξω ε, τώρα διαφάνειες. Ασχολούμαστε τώρα ε, με την εξυπηρέτηση ε, των πελατών μας και με την αλλαγή κάπως στην ενεργειακή πολιτική και νοοτροπία στη Γερμανία. Οπότε δεν θέλω να σας κουράσω με διαφάνειες, να σας πω μερικά πράγματα. Σας είπα ότι είμαστε μια μεσαία επιχείρηση, κλασική, ε, νερό, φυσικό αέριο, ε, ηλεκτρική ενέργεια και ανανεώσιμες φωτοβολταϊκά, βιομάζα, αιωλική ενέργεια κτλ. Περίπου ένα με 2% της παραγωγής φυσικού ε, ε, αερίου ηλεκτρικής ενέργειας είναι δική μας. Δεν ναι. είμαστε η δεν είμαστε μεγάλες εταιρείες ηλεκτρισμού, είμαστε λίγο παρακάτω. Ε, και έχουμε και εγκαταστάσεις που έχουμε συνδυασμένη παραγωγή ενέργειας και θερμότητας με τηλεθερμία και τηλεθερμασία και νοικοκυριών και δημοσίων κτηρίων ε, και ταυτόχρονα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη μείωση λοιπόν ε, του διεξουδίου του άνθρακα, μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και τις πράσινες θέσεις απασχόλησης. Εκεί δεν έχουμε άσπρο μαύρο, δεν έχουμε σωστό και λάθος. Είναι ένα σύνολο ε, μέτρων που μπορεί κανείς να πάει, μια δέσμη μέτρων για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, για τη μεγαλύτερη ε, συμμετοχή ανανεώσιμης ενέργειας. Όλα αυτά έχουν και ένα τίμημα, έτσι. Ε, μπορεί τελικά να είναι θετικά ή αρνητικά. Κάποιοι θα βρουν και αρνητικά. Δηλαδή, Τα αρνητικά μέτρα είναι μέτρα που δεν χρειάζονται χρήματα ή που αποδίδουν από μόνα τους, αυτό χρηματοδούνται, αλλά ε, αυτό δεν είναι πάντα ευπρόσδεκτο γιατί αλλάζει νοοτροπίες, ε, τακτικές και πρακτικές. Ε, βέβαια, για κάποια άλλα μέτρα χρειάζονται επενδύσεις ε, ο καλύτερος τρόπος συνήθως είναι διανόμου, να είναι υποχρεωμένος κανείς, αλλά και από εθελοντικές ε, ε, κινήσεις της βιομηχανίας με ίδιες πρωτοβουλίες που είναι και μια κίνηση marketing. Τώρα στη Γερμανία βγήκε ένα φυρμάνι, moratorium να, να μειωθεί η πυρηνική ενέργεια. Ε, βέβαια, ο προϋπολογισμός ε, είναι δεδομένος και υπάρχει οροφή λόγω της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. και θα επιστρέψουμε στη θερμοηλεκτρική ενέργεια, αν εγκαταλείψουμε την πυρηνική. σε ό,τι αφορά τους ευφύς μετρητές, τα, ρολόγια του ηλεκτρικού, να σας πω, εδώ εν παρόδο, ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε τίποτα θαύματα εξοικονόμησης ενέργειας ή ε, μετατόπιση από τις ώρες μεγάλης κατανάλωσης σε ώρες μικρής κατανάλωσης. Απλώς θα πρέπει να μάθουμε ε, ορισμένες συσκευές να τις χρησιμοποιούμε άλλη ώρα. Τις ειδήσει έτσι κι αλλιώς θα τις δούμε στις 8 ώρα το βράδυ, στις 9. Δεν πρέπει να αλλάξει η τηλεόραση. Ε, αλλά μπορείτε ας πούμε το στεγνοτήριο να το βάλετε το βράδυ, αν έχετε στεγνοτήριο. Ε, πλυντήριο, ε, πλυντήριο πιάτων, ε, ηλεκτρική σκούπα μπορούμε να αλλάξουμε ώρε που τι χρησιμοποιούμε, αλλά την τηλεόραση ή το φούρνο θα φάμε την ώρα που τρώμε και θα δούμε τι εκπομπέ που βλέπουμε σε συγκεκριμένε ώρε. Και μάλιστα όχι όλοι, μόνο εκείνοι που έχουν συνειδητοποιήσει και είναι ε, ενεργοί πολίτε ας πούμε. Και στην αρχή όταν είναι μόδα η συνείδηση είναι μεγάλη, αλλά σιγά σιγά εξατμίζεται. Μια φορά το χρόνο όταν έρχεται ο λογαριασμό για όλο το έτος, τότε ε, υπάρχει θυμός εκνευρισμός και μετά το ξεχνάμε. Λοιπόν, σε περίπτωση που πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, θα οξύνουμε, θα κάνουμε πιο αυστηρούς τους στόχους για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Ωραία, αλλά σε ποιο τομέα θα γίνει αυτό, στα νοικοκυριά. Όχι, αυτό δεν είναι δημοφιλές, διότι ε, πρέπει να επανεκλεγείς όταν είσαι πολιτικός. Στις μεταφορές, στις συγκοινωνίες, στη Γερμανία είναι δύσκολο αυτό. Βάλαμε μια ποσόστοση εθανόλης στη βενζίνη ή πιο εύκολο είναι να μειώσεις ε, το διοξίδιο του άνθρακα ε, στις εταιρείε, στις μεγάλες βιομηχανίες που καταναλώνουν πολύ και παράγουν διοξίδιο του άνθρακα, στη βαριά βιομηχανία, στο χάλιβα και σε μεγάλα εργοστάσια. Αυτό γίνεται, αλλά έχει και επιπτώσεις. Είναι πιο ακριβή η παραγωγή ενέργειας από ρηκτά καύσιμα και κοστίζει και περισσότερο ε, και σε εμά, αλλά αυτό το κόστος θα το μετακυλήσουμε στο τελικό χρήστη. Ε, που δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Γιατί είμαστε αγγελοφόροι κακών ειδήσεων και δεν μας αρέσει. Και δεν ισχύει ένα αξίωμα τη πολιτική. ότι τα πάντα γίνονται, αλλά τα πάντα έχουν επιπτώσεις. Από πλευράς εθνική οικονομίας γενικότερα, αν θέλουμε να το δούμε, εντάξει. Εμένα δεν θα με ενθουσίαζε κάτι τέτοιο. Ας πούμε ότι εφαρμόζεται, τι να κάνουμε. Αλλά αν το εφαρμόσουμε τότε με τρόπο που να μην ε, οδηγεί σε απόρριψη και σε... Παράδειγμα, η τρίτη περίοδος μορίας εκπομπών από το 2013 και μετά, εκείνοι που παράγουν θερμότητα, παίρνουν λιγότερα πιστοποιητικά για το διοξίδιο του άνθρακα. Ενώ εκείνοι που έχουν μικρή παραγωγή με ένα μικρό λέβητα ή με ένα μικρό ε, καζάνι, ξέρω εγώ, σε μια πολύ περιορισμένη ποσότητα, δεν δικαιούνται πιστοποιητικό. Εδώ ε, όμως αυτό οδηγεί σε στρεβλώσεις υπάρχουν πόλεις όπως είναι Βρυξέλλες, η κολονία που είμαστε εμείς, ε, με κεντρική παραγωγή θέρμανσης είμαστε σε συγκριτικό μειονέκτημα από τους μικρούς παραγωγούς πολυτοπικούς. Και όποιος θέλει να μειώνει το διοξίδιο του άνθρακα θα πρέπει να έχει μια κρίσιμη μάζα για να μπορεί ουσιαστικά να μειωθεί το διοξίδιο του άνθρακα. Να, έχει ένα μέγεθος ο παραγωγός. Τώρα για τους ευφύς μετρητές δεν ξέρω πώς ε, ορίζεται αυτό και πώς θα γίνει. Αυτά. Ήθελα να σας πω έτσι κάποια σκόρπια σχόλια και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα εγώ έχω το άχαρο έργο να κοιτάω το ρολόι. Δεν είναι μόνο η ενεργειακή απόδοση, είναι και η χρονική. Χωρίς να αφλιαρώ, θέλω να δώσω λόγο στον επόμενο μιλητή που είναι ο κύριος Ρεμί Γκρουέ από την ΕΒΕΑ που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αεολική Ενέργεια και θα μας πει ποια βήματα πρέπει να γίνουν και από πλευράς υποδομής τι πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε να φτάσουμε και στους στόχους που συζητάμε αυτό το καιρό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Γκρότε, θα μιλήσω αγγλικά. Από ό,τι φαίνεται κυκλοφόρησε η παρουσίασή μου. Ε, ε, αγγλικά είπα, γιατί τα λέω γερμανικά. εκπροσωπούμε τους κατασκευαστές τουρμπινών αιωλικής ενέργειας αλλά και όλων των υπολείπων εγκαταστάσεων που χρειάζονται για την παραγωγή της. Θα σας πω πού βρισκόμαστε τα τελευταία 10 χρόνια και πού αναμένουμε να φτάσουμε τα επόμενα 10. Συνεχώς αυξάνονται οι δυνατότητες θεολικής ενέργειας στην Ένωση Μέχρι το 20 υπολογίζουμε να φτάσουμε στην παραγωγή 230 κιλοβατορών ανά ανά κάτοικο. Εκρηκτική αύξηση λοιπόν. Α, Εδώ θέλω να σας δείξω ότι η ολική ενέργεια είναι ήδη σημαντικό ποσοστό της συνολικής παραγωγής ενέργειας σε πολλές χώρες. Στη Δανία ιδίω 24%, Πορτογαλία, Ισπανία περίπου 15%, Γερμανία και Ιρλανδία προς το 10% και ο μέσος όρος της Ένωσης 5,3%. Οι υπόλοιπες χώρες ε, επίσης ε, κάνουν μαζικές παραγγελίες. Ποιες είναι, ποια είναι τα μακροοικονομικά ωφέλη. Ενεργειακή ασφάλεια, εξοικονομήσεις από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, μείωση του κόστους για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών γιατί δεν υπάρχει καθόλου εκπομπή διοξιδίου από την αιωλική ενέργεια ε, δυνατότητες εξαγωγών, δημιουργία θέσεων εργασίας, 188.000 το 2010 μέχρι και 450.000 το 2020 και τέλος όπως είπε και ο προηγούμενος για να μην αυξηθεί το κόστος της παραγωγής ενέργειας λόγω της πολέμησης του διοξιδίου ορίστε μια λύση η αιωλική εδώ βλέπετε το merit order effect που λέμε γιατί η αιωλική ενέργεια μειώνει τις τιμές της ενεργείας και τις εκπομπές. Η καμπύλη αυτή βασίζεται στο περιθωριακό κόστος, όχι στην επένδυση. Δείχνει απλώς πώς δουλεύει η αγορά. Η αιωλική και άλλες ανανεώσιμες πηγές ε, γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Κάτω αριστερά Βλέπετε ότι γράφει παραπάνω αΐρ, Ενώ δεξιά γίνεται η τομή με την καμπύλη της ζήτησης. Σε μερικές χώρες έχει υπολογιστεί ότι μειώνονται οι τιμές κατά ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο που απέτησαν οι επενδύσεις. Πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα ότι η αιωλική ενέργεια μπορεί να είναι και φτηνότερη από τις άλλες. Τώρα, εάν είναι λύση κλειδί για τις κλιματολογικές αλλαγές, μέχρι το 2010 μειώσαμε εκπομπή κατά 126 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου αλλά μέχρι το 2020 αναμένουμε να αυξηθεί αυτό στους 342, στα 342 εκατομμύρια ισοδυνάμου, 30% δηλαδή. Δεν είναι δύσκολο να φτάσουμε στο στόχο αυτό του 30%. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές είναι οι πρωτοπόροι στον κόσμο στην κατασκευή τουρμπινών. 96% παγκοσμίω. Τεράστιο ποσοστό. Στη ΣΥΠΑ και την Κίνα όμως επίσης είναι οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, έχουν μεγάλο μερίδιο. Το μεγαλύτερο μερίδιο είναι εντόπιον κατασκευαστών, αλλά οι Ευρωπαίοι έχουν μεγαλύτερο μερίδιο από όλους τους μη ντόπιου κατασκευαστές. Ο κύριος Γκέμπελς έφυγε, αλλά θα ήθελα να αμφισβητήσω αυτό που είπε ότι η Κίνα έχει γίνει ο μεγαλύτερος εξαγωγεύς εναλλακτικών ενεργειών. Η Ένωση είναι. Η άλλη πλευρά της τεχνολογίας βέβαια είναι ο ηγετικός ρόλος που πρέπει να παίζουμε τεχνολογικά. Στην Ευρώπη έχουμε τεχνογνωσία, υλικά, οι δυνατότητες έρευνας, πανεπιστήμια και δίκτυα και η εμπειρία μας εκτός Ένωσης είναι πολύ μεγάλη. Επίσης, εδώ και 15 χρόνια υπάρχει, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και άλλες χώρες επενδύουν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ταϊβάν. Έχουμε λοιπόν αυτό το τεχνολογικό όφελος, αλλά υπάρχουν και με σοβαροί ανταγωνιστές. Η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή φιλόδοξα προγράμματα ανανεωσίμων. Η Κίνα με το νέο πενταετές της σχέδιο προσθέτει 70 γιγαβάτ δυνατότητα. Ο Δε Ομπάμα στο λόγο του για την κατάσταση της Ένωσης είπε ότι θα στηρίξει περαιτέρω αιωλική ενέργεια και το μέγεθος των αγορών αυτών τους βοηθάει. Η ευρωπαϊκή αγορά έχει περίπου τις ίδιες διαστάσεις με των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ η κινέζικη είναι πολύ μεγαλύτερη και ανάλογες επενδύσεις γίνονται όπως βλέπετε εδώ. Πρέπει οι Ευρωπαίοι επενδυτές να τύχουν κάποιας ενθάρρυνσης για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Φαίνεται ότι η κρίση έπληξε και τον τομέα αυτόν η τιμή του διοξιδίου του άνθρακα δεν ενθαρρύνει τα πράγματα. Δύο λύσεις υπάρχουν ή να αυξήσουμε τις δυνατότητες μας αμέσως στο 30% ή να έχουμε περισσότερες επιχορηγήσεις. Η βαριά βιομηχανία βέβαια έχει άδειε που επιτρέπουν να περάσουμε στο το κόστος για την αντιμετώπιση του οξυδίου 100% στους καταναλωτές. Οι επενδύσεις στις υποδομές δικτύων θα ήταν ωφέλιμες για όλους, θα μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των υπαρχόντων συστημάτων, αλλά επίσης χρειάζονται περισσότερες διαμεθοριακές συνδέσεις για να μπορεί να χρησιμοποιείται η ελληνική ενέργεια όποτε και όταν χρειάζεται, αλλά και να διασφαλίζει την ασφάλεια των προμηθειών. Εδώ βλέπετε ότι οι επενδύσεις που χρειάζονται για τις ανανεώσιμες είναι οι χαμηλότερες από το τρία είδη. Και τώρα τα συμπεράσματα. Χρειάζεται παγκοσμίω να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου και ή θα επενδύσουμε σήμερα στα εναλλακτικά προϊόντα ή θα περιμένουμε να αγοράσουμε κάποιο άλλο. Η εφόσον η Ένωση έχει τεχνολογικό βασικό προτέρημα εδώ στις ανανεώσιμες. Χρειάζεται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που να αντιμετωπίσει, να πετύχει αυτόν τον στόχο του 30, της μείωσης κατά 30% και πρέπει να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα καινοτομιών. Και ήδη από τώρα να αρχίσουμε να συζητάμε τους στόχους για τους ανανεώσιμες κατά 30%. Σας κατευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δέκα λεπτά ακριβώς, με το ρολόι. Πολύ ενδιαφέροντα και τα στοιχεία που μας είπατε. Για να φτάσουμε στους στόχους μας. Επόμενος ομιλητής τώρα είναι ο κύριος Χουνέν από την UMP, διευθυντής. Έχετε το λόγο και εσείς για 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές. Θα κάνω μια σύντομη επισκόπηση για το πώς αντιλαμβάνονται τη συζήτηση και η παραγωγή ενέργειας και οι μεγαλύτεροι χρήστες ενέργειας. Η UPM είναι μια ε, πανευρωπαϊκή, ε, ένας πανευρωπαϊκός όμιλος που εδρεύει στη Φιλανδία ε, για την υλοτομία και έχουμε συνεργασία με τους μεγαλύτερους εταίρους στην αγορά. Βέβαια κυρίως έχουμε το 70% των εισόδων από τη χάρτοβιομηχανία και θα επικεντρωθώ κυρίως σε αυτή την πτυχή στην παρουσίασή μου. Βέβαια, δημιουργούμε και νέες ευκαιρίες, ανάπτυξη βιοκαυσίμων, για παράδειγμα, και ε, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση από τη Γαλλία και Φιλανδία στο NER 300 και έχουμε και πολλές, ε, πολλά εργοστάσια ε, βιοχημικά και RFID. Είμαστε μια εταιρεία με 70% του τζίρου μας να προέρχεται από την Ευρώπη, αλλά έχουμε δραστηριότητες και στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Νότια Αμερική. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, νομίζω η θέση μας είναι καλή, γιατί μπορούμε να αξιολογήσουμε πού μπορούμε να επενδύσουμε και πού είναι πιο αποδοτικές οι επενδύσεις της εταιρείας μας. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, Έχουμε 3.000 ΜΒ ε, δυναμικό παραγωγής. Είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας στη Φιλανδία και καταναλώνουμε 12% του, της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της Φιλανδίας. Παράγουμε 30% των ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας και 1% των συνολικών εκπομπών ε, διοξίδιου του άνθρακα. Είμαστε δηλαδή μια εταιρεία ε, που ε, καταναλώνει πολλή ενέργεια, αλλά δεν παράγει πολλά καυσαέρια. Και το 20% της ε, παραγωγής ενέργειας προέρχεται από δεύτερες πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είχαμε σημαντικές επενδύσεις και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε μερικά παράδειγμα. Έχουμε ε, το μεγαλύτερο εργοστάσιο στον κόσμο που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είμαστε η δεύτερη, μεγαλύτερη, το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο που παραγωγεί ενέργεια με βιομάζα στην Ευρώπη. Εδώ μιλούμε ταυτόχρονα και για αξιονόμηση και για ενεργειακή απόδοση, για διαρροή άνθρακα, για κλιματικές πολιτικές. Η ενεργειακή απόδοση της, ήταν αναπόσπαστο τμήμα ανέκαθεν της βιομηχανίας μας και από την αρχή αναλάβαμε κάποιες πρωτοβουλίες σχετικά γιατί η λογική της επιχείρησής μας είναι ε, να κάνουμε καλύτερη αξιοποίηση και των πρώτων υλών και οποιασδήποτε άλλη πηγή. Θέλουμε απόδοση, αποτελεσματικότητα των προϊόντων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούμε και από το 1990 η κατανάλωση ηλεκτρισμού ανατόνου χάρτου έχει μειωθεί γύρω στο 40%. Από το 97 μάλιστα και μετά μειώθηκε κατά 23%. Την τελευταία διετία εφαρμόσαμε στη χαρτοβιομηχανία μας μία πρωτοβουλία όπου όλο το προσωπικό συμμετείχε σε αυτή την πρωτοβουλία και ξοδέψαμε 9 εκατομμύρια. Ε, λάβαμε 140 ιδέες και 9 εκατομμύρια ε, ξοδέψαμε, εξοικονομήσαμε 27, 25 εκατομμύρια και 7 εκατομμύρια τόνους ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Φυσικά θα πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, πιο αποδοτικοί μάλλον, να εξοικονομούμε περισσότερη ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε και την ανταγωνιστικότητά μας. Και φυσικά είμαστε από τους ε, καλύτερους παραγούς ό,τι αφορά το κόστος και την αποδοτικότητά μας. Η διαφάνεια αυτή περιγράφει τις νανοίνες που είναι βασικός τομέας έρευνας. Βρισκόμαστε πραγματικά σε ένα σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά αυτή την καινοτομία και υπάρχουν πολλές αλληλεπιδρούμενες, αλληλένδετες πολιτικές προσπαθούμε να δούμε το συνολικό αντίκτυπο όλων αυτών των πολιτικών. Η χαρτοβιομηχανία υπόκειται τεράστιες πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία. Μάλιστα είχαμε για πολλά χρόνια μια πτωτική πορεία των τιμών και σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες, ε, ειδικά τον ηλεκτρισμό, η πορεία είναι ανωδική. Οπότε για να είμαστε πραγματικά ανταγωνιστικοί πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί και για να αξιοποιούμε καλύτερα τι πηγέ μα. Υπάρχει και δερμή ανταγωνισμό εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέε επενδύσει στη χαρτοβιομηχανία έγιναν κυρίω στην Κίνα και την Νότια Αμερική. Πώ θα εξασφαλίσουμε λοιπόν τη βιωσιμότητα του κλάδου, πώ θα διαφυλάξουμε την ανταγωνιστικότητά μα, πώ θα κρατήσουμε ανθούσα τη βιομηχανία μα και θα προστατεύσουμε τι θέσει απασχόλησή μα. Θα ήθελα να σας επισημάνω επίσης ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ιδιάζουσα κατάσταση ό,τι αφορά τα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί ε, επειδή η χαρτοβιομηχανία στηρίζεται στα δάση, στην υλοτομία, παράγουμε με ανανεώσιμες ενέργειες, αλλά και εκεί ε, έχουμε τεράστιες πιέσεις στις πρώτες ύλες. Γιατί υπάρχει χρήση του ξύλου για την παραγωγή ενέργειας και πολλές φορές ε, οι πυρκαγιές επίσης μας ε, επηρεάζουν πολύ αρνητικά. Έχουμε εδώ ένα τριπλό κίνδυνο σε ό,τι αφορά τις ε, συναφείς με την ενέργεια πολιτικές που εξετάζουμε σήμερα. Υπάρχει καταρχήν ο αντίκτυπος του κόστους των αδειών εκπομπών το αυξανόμενο κόστος του ηλεκτρισμού, αλλά υπάρχει και το κόστος ε, της πρώτης ύλη, του ξύλου δηλαδή για μας. Και αυτός ο συνδυασμός μας φέρνει σε δυσάρεστη θέση σε ό,τι αφορά την επιλογή των επενδύσεών μας. Πρόσφατα αναγγείλαμε τις ε, προτεραιότητες μας στις επενδύσεις. μόνο ένα προτεραιότητα είναι οι επενδύσεις σε, Ευρωπαϊκή. Ε, αποτελεσματικότητα και οικονομική απόδοση. Επίσης, ε, σε συνδυασμένες ε, παραγωγές θερμότητας και ηλεκτρισμού και μας ενδιαφέρει φυσικά ο, η σχέση κόστος-οφέλους και αγοράσαμε με 900 εκατομμύρια ευρώ μια άλλη χαρτοβιομηχανία στην Ευρώπη και μάλιστα η συγχώνευση που εξετάζεται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζουμε ότι θα μας επιτρέψει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στον κλάδο. Όπως σας είπα, εξετάζουμε και κάποια προγράμματα βιοκαυσίμων στη Γαλλία και Φιλανδία. Έχουμε και μια άλλη επένδυση που σχεδιάζουμε 500 εκατομμυρίων στη χαρτοβιομηχανία της Κίνας και πάνω από ένα δις ε, ε, επενδύσεις, επενδυτικά σχέδια στο νότιο ημισφαίριο. Πρόκειται για περίπλοκες επενδυτικές αποφάσεις. Πάντως ε, μπορώ να πω σήμερα δεν μπορώ να πω με ακρίβεια τι αντίκτυπο θα έχει η, μία, η α ή β πολιτική. Πάντως γενικά για να εξασφαλίσουμε τη θέση της αβιομηχανίας στην Ευρώπη είναι το σύνολο των προϋποθέσεων και των συνθήκων να τίνουν υπερμίας ανταγωνιστικότητας. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα θέλαμε να δούμε μια πιο βιώσιμη οικονομία, πιο φιλοπεριβαλλοντική και επίσης ο ρόλος των βιοχημικών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ανανεώσιμων πρώτων υλών. Ο ρόλος τους θα αυξηθεί στο μέλλον όλο και περισσότερο. Και ειδικά για μας τη χαρτοβιομηχανία Χρησιμοποιούμε βιοδηληστήρια που χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πρώτες ύλε σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό και είμαστε σε θέση να προωθήσουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Πάντως, για να γίνουμε πραγματικά ο γίγαντας των φιλοπεριβαλλοντικών χημικών και των βιοκαυσίμων, χρειαζόμαστε ρευστό και χρειαζόμαστε εύρωστες επιχειρήσεις και ανταγωνιστικές φυσικά επιχειρήσεις που θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν αυτό το βήμα. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τις, τη συζήτηση για τις πολιτικές, το μήνυμά μας είναι απλό. Εμείς, αυτό που θέλουν οι επιχειρήσεις είναι προβλεψιμότητα. Η στρατηγική του 2020 σε ό,τι αφορά τι επενδυτικές μα αποφάσει, είναι πολύ κοντά. Το 2020 είναι πολύ κοντινό ορίζοντας. Χρειαζόμαστε όμως ένα σταθερό επενδυτικό πλαίσιο που δεν θα αλλάζει κάθε τρει και λίγο, γιατί μία αλλαγή δημιουργεί αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα σίγουρα δεν μας ικανοποιεί. Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάνν Χούνεν, και για την παρουσίαση και για την απεικόνηση. Ήταν πάρα πολύ ε, εύγλωτη μία από τις τελευταίες διαφάνειες. Έχει έρθει η ώρα της συζήτησης τώρα. Η Λένα Εκ πρώτη και μετά βλέπουμε. Είναι από τις καλύτερες εταιρείες παγκοσμίω ως προς τη βαθμολογία της εταιρείας σας και αξίζει ε, αυτή την κατάταξη της UPM Κείμενε. Πώς ε, θα ε, εξισορροπήσετε την παραγωγή με το εισόδημα. Εσείς είστε ηγέτες στην κατάταξη. Πώς θα μπορούσατε να μεταφέρετε την εμπειρία σας στην Ευρώπη στο σύστημα συνδυασμένης παραγωγής. Πώς μπορεί αυτό να μεταφερθεί στην Ευρώπη, το παράδειγμά σας. Ευχαριστώ. Η Αντίτ Χερτσόκ, την επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω για την αιωλική ενέργεια. Για την ανταγωνιστικότητα. Έχουμε μεγάλη τεχνογνωσία στην Ευρώπη, αλλά σιγά σιγά χάνεται με το χρόνο. Το θεωρείτε πρόβλημα, θέλετε να το συζητήσουμε, πρέπει να το συζητήσουμε πώς διαχειρίζεται η Ευρώπη τη γνώση της. Ιδιαίτερα τη βιομηχανική και τις εφευρέσεις είναι από ό,τι φαίνεται αξία και συγκριτικό πλεονέκτημα, αν μπορεί η Ευρώπη να το κάνει. Αλλά πόσο μπορούμε ακόμα να εξασφαλίσουμε αυτό και να καλύπτουμε την απόσταση. Αλλιώς, εμείς έχουμε στόχους της λισαβόνα. αλλά αν τους στόχους αυτούς δεν τους αξιοποιήσουμε, δεν είναι πλέον αξία, είναι κόστος, είναι μειονέκτημα. Ε, ρωτώ όλους, αλλά εσείς κυρίω από την αιωλική ενέργεια το αναφέρατε περισσότερο. Ευχαριστώ. Δύο συνάδελφοι λοιπόν ρώτησαν. Θα πρότεινα να απαντήσετε πρώτα ο κύριος ε, Γιάνχουνεν και μετά ε, ο κύριος Κρούετ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και για τις ε, παρατηρήσεις σας. Είναι ευκαιρία, βεβαίως, ε, στις ε, βορειοευρωπαϊκές χώρες η συνδυασμένη παραγωγή ενέργειας και θερμότητας, αυτό το CHP, έχει κερδίσει έδαφος για λόγους ευνόητους, ε, κλιματολογικούς. Και ε, η θερμότητα που παράγουμε διοχετεύεται στο δίκτυο θέρμανσης στο αστικό. Είναι πάρα πολύ κοινή, ε, πρακτική και συνηθισμένη και στη Σουηδία και στη Φινλανδία. Σε άλλα μέρη της Ευρώπης δεν χρειάζεται τόσο πολύ ε, αυτή η θέρμανση. Το καλοκαίρι σταματάει και στη Φιλανδία, αλλά εμάς είναι η ανάγκη μας εκ των πραγμάτων. Τώρα, αν μεταφέρεται αυτό στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, απομένουμε να το δούμε. Έχουμε επενδύσει στην Αυστρία, στη Γερμανία, στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο σε τέτοια εργοστάσια συνδυασμένη παραγωγή θερμότητα και ενέργεια. Ε, απειλή βλέπω και πάλι από πλευρά των δασών. Εμείς παράγουμε κάποια προϊόντα και τα υποπροϊόντα τα χρησιμοποιούμε για παραγωγή ενέργειας. Αλλιώ, εάν υπερισχύσει πολύ η παραγωγή θερμότητα και ενέργεια. αυτό θα είναι βάρο των βασικών μα προϊόντων, που είναι προϊόντα χάρτου. Ναι, μπορεί να υπάρχουν και απόβλητα που να χρησιμοποιούνται σε αυτή την προσπάθεια, βεβαίω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρουέτ. Στα αγγλικά... Μπερδεύομαι, πάω να μιλήσω γερμανικά, αλλά πρέπει να μιλάω αγγλικά. Πώς διατηρούμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Καταλαβαίνουμε ότι φτάσαμε εδώ με το 1% της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για έρευνα για προβλήματα για τα καινοτομίας. Το καταφέραμε λοιπόν αυτό με 1% του ενεργειακού προϋπολογισμού να πηγαίνει στην έρευνα. Υπάρχει βεβαίω σαφή ανάγκη συνέχισή ε, της δημόσιας χρηματοδότησης στην έρευνα και την καινοτομία. Με ενδιαφέρει αυτό. Νομίζω ότι είναι ε, η πρόβλεψή σας 6 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι δεν είναι. Για την αιωλική ενέργεια. Για να κοιτάξουμε ποιες είναι οι επόμενες τεχνολογίες που μπορούμε να παράγουμε, να αναπτύξουμε. Αυτό θα είναι πάρα πολύ κλειδί <laughs> για το μέλλον. για να ξέρουμε πού θέλει να καταταγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την προσπάθεια και χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις ιδιωτικές από τις εταιρείε. Δεν είναι ιδιωτική χρήματο, ε, δημόσια, συγγνώμη. Το 95% των offshore ανεμογεννητριών στη θάλασσα είναι ιδιωτικές επενδύσεις. Χρειαζόμαστε και στόχους και ε, χρήματα. Τελευταία ερώτηση. Ισά του χάσει. Για να περάσουμε στο επόμενο πάνελ, σιγά σιγά. Γιατί και πάλι σας είπα έχω το άχαρο, ε, ε, αχάριστο καθήκον να κοιτάω το ρολόι. Okay, thank you very much. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τα σχόλια από, εκπρόσωπ, από εκπροσώπους ε, επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ό,τι αφορά το μελλοντικό πενταετές ενεργειακό πρόγραμμα της Κίνας. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι πιθανό η Κίνα όχι μόνο από άποψη όγκου παραγωγής αλλά και από άποψη τεχνολογίας είναι πιθανό να κινηθεί πολύ ταχύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μας ξεπεράσει και στην τεχνολογία. Τι συμπεράσματα μπορούμε να συνάγουμε από τις φιλοδοξίες της Κίνας για τη χρήση νέων τεχνολογιών. Νομίζω είναι μια εμπειρία που αφορά τώρα το κλάδο των φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη. Mm. Μέχρι τώρα οι Γερμανοί, οι Άπωνες και οι Ευρωπαίοι παραγωγοί ε, ήταν ηγετικοί στον κόσμο. Τώρα μας ξεπέρασε η Κίνα mm. που έχει καταλάβει πολύ μεγάλα μερίδια της αγοράς και για λόγους τιμών. Και από το 2009 έχει γεμίσει η Γερμανία φωτοβολταϊκά και γίνεται μεγάλη φασαρία πώς το καταφέραμε αυτά, περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ε, μισθή, σίγουρα είναι μια δέσμη ε, παραγόντων. Δεν ξέρω αν αυτό λειτουργεί και σε άλλες τεχνολογίες και αν μας βγαίνει εξίσωση. Ε, δεν ξέρω. Ε, θα σας πει και ο συνάδελφος για την νεολική ενέργεια. Χρειάζεται προσοχή όμως να μην χάσουμε το τρένο. Εξάλλου δεν έχουμε και τόσες πρώτες ύλε στην Ευρώπη. Και θα μας ξεπερνάνε άλλοι που θα έχουν έτσι τέτοια επιθετική πολιτική. Να πω κι εγώ δύο λόγια. Αυτό που συνέβη εν μέρος ε, ε, σε αυτή την ενέργεια, την ενέργεια δεν μπορεί να συμβεί παντού. Ας πούμε για τις, ε, για τις ανεμογεννήτριες το ίδιο κόστος έχει να την παράγει στην Κίνα, το ίδιο να το παράγει και στην Ευρώπη. Ε, αν δούμε μάλλον και, το κόστος εξαγωγής από την Κίνα στην Ευρώπη δεν είναι πάρα πολύ ε, αποδοτικό. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε εργοστάσια στην Ευρώπη. Μπορούμε να εξάγουμε στους γείτονές μας, αλλά όχι πολύ μακρύτερα. Όπως σας είπα, η κινέζικη αγορά ήταν πολύ ισχυρή σε τιμές, σε, σε φθηνά προϊόντα. Εμείς είμαστε πιο ισχυροί σε προϊόντα, ε, προϊόντα ψηλής ποιότητας, με μεγάλη καινοτομία, με μεγάλη ποιότητα. Έχουμε στόχους, έχουμε ε, κίνητρα και για τη χρηματοδότηση της έρευνας. Αλλιώς θα, θα πρέπει να ζητάμε να κλείσουν τα σύνορα για να μην μας κατακλείσουν τα κινέζικα προϊόντα. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και για τις ερωτήσεις που απαντήσατε. Ε, βλέπουμε ότι ο δρόμος δεν είναι εύκολος, ο οποίο έχουμε διαλέξει, είτε είναι 20% είτε 30% και πάλι σας ευχαριστώ που ήρθατε, αλλά και για τις παρουσιάσεις σας, πολύ ε, καλές. Ε, παρακαλώ να έρθει το επόμενο πάνελ που αφορά την καινοτομία και την έρευνα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Χρειάζεται προσοχή και πάλι εδώ να μην χάσουμε το τρένο της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας και ε, περιμένω να ακούσω τις τοποθετήσεις ε, των εμπειρογνωμόνων. Έχουμε τον κύριο Λαμπερτερή που είναι Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής ε, Πλατφόρμας Τεχνολογίας του Χάλιβα και τον κύριο Νίλσεν που είναι ο Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην εταιρεία Novozim, αν σωστά το αναφέρω, αλλιώ παρακαλώ να με διορθώσετε. Και θα πρότεινα να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Λαμπερτερή Remote Control. Das ist einmal, dass die Technik freigeschaltet wird, dass wir... Για να ετοιμάσουμε και τα θέματα τα τεχνολογικά και τα διαδικαστικά και έχετε μέσα στο λόγο κύριε Λαμπερτερίν. Et dans son agenda de recherche stratégique, Κοιτάξτε, στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής προσέγγισης, ένα από τα κυριότερα είναι, θέματα είναι η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος από τη χαλιβουργία. Pour produire l'acier, il existe deux familles de procédés. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι. Πρώτον, η χρησιμοποίηση του συντηρομεταλλεύματος από τις υψικαμίνους για τη δημιουργία υγρού χάλιβα ή η ανακύκλωση του σιδηρομεταλλεύματος. Στην Ευρώπη παράγονται περίπου, στην Ευρώπη των 27, 200 εκατομμύρια τόνοι το χρόνο, 60% από σιδηρομετάλλευμα και τις υψηκαμίνους και 40% από την ανακύκλωση με ηλεκτρικούς φούρνους. Από, ηλεκτρι... από ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές η μέθοδος του σιδηρομεταλλεύματος απαιτεί πολύ περισσότερη ενέργεια και άρα εκπομπή διοξιδίου λόγω της ζήτησης από τη χημιομηχανία. Κατά μέσο όρο μπορεί κανείς να πει ότι αν συμπεριλάβουμε την εκπομπή διοξιδίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκπέμπονται τέσσερις φορές λιγότερα χαμηλότεροι όγκοι από τη δεύτερη μέθοδο διοξιδίου παρά από την πρώτη. Τα τελευταία 40 χρόνια μειώσαμε κατά 50% την κατανάλωση ενέργειας και άρα και τις εκπομπές διοξιδίου. Σε σύγκριση με αυτά που είπαμε το πρωί θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σύνδεση μεταξύ ενεργειακής αποδοτικότητας και εκπομπής διοξιδίου. Και αυτό το πετύχαμε πρώτον διότι αυξήθηκε η ανακύκλωση του μεταλλεύματος υπήρξε, σημειώθηκαν πρόοδοι στην, στον τρόπο παραγωγής του χάλιβα και βελτιώθηκε η αποδοτικότητα της παραγωγής του. Σήμερα θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει στα τεχνολογικά όρια της παραγωγής αυτής και με την υπάρχουσα τεχνολογία έχουμε σχεδόν ίδια παραγωγή με τη θερμοδυναμική μέθοδο, με την υπάρχουσα λέω πάντα τεχνολογία. Τι προκλήσεις αντιμετωπίζουμε για το μέλλον. Απ' τη μία για να μειωθούν οι εκπομπέ διοξιδίου στην παραγωγή χάλιβα πρέπει να αυξηθεί η ανακύκλωση του μεταλλεύματος, να υπάρξουν ανταλλαγές βελτίστων πρακουτικών και να καταργηθούν οι απαρχαιωμένες μονάδες. Οι λύσεις λοιπόν για το χάλιβα μπορεί να υπάρξουν μέσω της εξοικονόμησης της παραγωγής λιγότερου διοξιδίου του άνθρακος στη διαδικασία παραγωγής του χάλιβα. Το 4 αρχίσαμε το πρόγραμμα ULCOS, Ultra Low, Carbon Steel Making Now και έτσι μπορέσαμε να καταργήσουμε τέσσερις μεθόδους παραγωγής απαρχαιωμένες και ταυτίσαμε εκεί τις τέσσερις αυτές κατηγορίες. Πρώτον, την ανακύκλωση του αερίου των υψηκαμίνων και τον διαχωρισμό του και την αποθήκευση του. Τα άλλα δύο θα τα πω μετά. Το ένα είναι μια εναλλακτική λύση για τις υψηκαμίνους, αντί για τις υψηκαμίνους. Και υπάρχει και η μέθοδος της ε, η ηλεκτρική μέθοδος με ηλεκτρόλυση. Ως προς το timeline έχουμε ταυτίσει ήδη τι πρέπει να γίνει μέχρι το 11 και έχουν τελειώσει τα πιλωτικά προγράμματα που έχουμε εγκρίνει. Φανταζόμαστε ότι αν πετύχουν αυτά τα πιλωτικά προγράμματα και τα πειραματικά τι αυτά θα μπορέσουμε μετά το 2020 να κάνουμε βιομηχανική παραγωγή. Εδώ βλέπετε την αποδοτικότητα ως προς την μη εκπομπή διοξιδίου των διαφόρων μεθόδων παραγωγής χάλιβα η μείωση κατά 50% του διοξιδίου, της εκπομπής διοξιδίου με την ανακύκλωση του αερίου και το CCS, δηλαδή το σύστημα αποθήκευσης. Το δεύτερο, η δεύτερη μέθοδος επιτρέπει κατά 4, 400% ε, μείωση. Μεγαλύτερη από το συνδυασμό των υψηκαμίνων και της ανακύκλωσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ε, εξαρτάται από τη χρήση που κάνουμε και αν θέλουμε να τα συνδυάσουμε όλα δηλαδή το διοξίδιο που χρειάζεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολό της τότε με τις σημερινές μεθόδους δεν υπάρχει, δεν έχουμε συμφέρον να το κάνουμε, δεν αποδίδει τίποτα. Αντίθετα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν διοξίδιο, θα ήταν πιο ενδιαφέρον. Le top guys recycling, on donc on prend le gaz de fourneau, on... Παίρνουμε λοιπόν εδώ σε αυτή τη μέθοδο το αέριο από τις υψηκαμίνους με συνολική μείωση της εκπομπής λόγω καλύτερης αποδοτικότητας και το διοξίδιο το αποθηκεύουμε υπογείως. Τώρα για αυτήν τη μέθοδο έχουμε καταθέσει πριν από ένα μήνα μία πατέντα που τη λέμε New Entrance Reserve Τα δικαιώματα εκπομπής λοιπόν κατά 300 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσουν 8 προγράμματα εναλλακτικά. Εφόσον εγκριθεί βέβαια το σχέδιο που υποβάλαμε. Θα πειραματιστούμε επίσης στο Eisenhüttenstadt στη Γερμανία τι δυνατότητες υπάρχουν ανακύκλωσης του διοξιδίου, ε, άλλες. Η δεύτερη μέθοδος, δεύτερη, τελείως καινούρια, είναι μείωση και τήξη. Δηλαδή χρησιμοποιείται απευθεία στο συνδρομετάλλευμα το διοξίδιο και το, ο άνθρακας και παρα, ε, εκπέμπεται λιγότερο διοξίδιο το οποίο όμως αποθηκεύεται μετά πιο εύκολα από το πρόγραμμα CCS Carbon Capture and Storage. Υπάρχει και εδώ ένα πειραματικό πρόγραμμα με στήριξη του, της Ολλανδικής κυβέρνησης το πρόγραμμα Χισάρνα που θα αρχίσει τον Απρίλιο 11 Βλέπετε εδώ τι ωραία φωτογραφίες Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Χάλιβας μπορεί επίσης να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου. Par co Πώς μέσω της χρησιμοποίησης του με αποδοτικότερο τρόπο γιατί εδώ υπάρχουν πολλές εφαρμογές στον ενεργειακό τομέα, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στις κατασκευές, στις οποίες όμως είναι δύσκολο να δώσουμε αριθμούς ως λόγους τουλάχιστον, γιατί υπάρχει το retrofitting που λέμε. Αυτό πώς να το υπολογίσουμε το retrofitting. Μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρχει παράγοντας 10 όμως. 10. Η παραγωγή χάλιβα στην Ευρώπη γενικά μείωσε κατά 50% τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και βελτίωσε κατά 50% την αποδοτικότητά της τα 40 τελευταία χρόνια. Ακόμα όμως μπορεί να γίνει και άλλη πρόοδος με την ανακύκλωση του μεταλλεύματος και τις καλύτερες εγκαταστάσεις. Η δραστική όμως μείωση των εκπομπών σημαίνει ότι πρέπει να πετύχουν πρώτα τα πειραματικά προγράμματα που αρχίζουν ήδη φέτος και θα αναδιπλωθούν σε 10 χρόνια. Αν πετύχουν και είναι και αποδοτικά οικονομικά, και γίνει αποδεκτό το σύστημα της αποθήκευσης του διοξιδίου, τότε θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους αυτές βιομηχανικά από το 20 και μετά. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ κύριε Λαμπερτερή. Πάρα πολύ ωραία τα είπατε. Ναι, ναι, ναι. Και ε, δείξατε ότι το CCS δεν είναι απαραίτητο μόνο για την παραγωγή ενέργειας, αλλά ε, και στη χαλιβουργία, όπου δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να μηδενιστεί η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, απολύτως. Εκεί λοιπόν ε, βρίσκει εφαρμογή και η δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Και επίσης μας αποδείξατε ότι υπάρχουν όρια από πλευράς φυσικής. Εννοώ τη φυσική την επιστήμη. Εγώ είμαι μηχανικός mm. και το κατάλαβα πάρα πολύ αυτό που είπατε. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Ε, περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ο κύριος Νίλσεν είναι έτοιμη και η παρουσίασή του στον υπολογιστή και μπορούμε να αρχίσουμε και μετά θα συζητήσουμε. Thank you and thank you for inviting me. Um, ευχαριστώ. Ε, που με καλέσατε να σας πω τι είναι η Novozymes. Είναι στη βιοτεχνολογία παγκόσμιος ηγέτης στα ένζημα για ε, ζωοτροφές, τρόφιμα, για είδη ένδυσης και στην έρευνα και στην ανάπτυξη είμαστε πρώτη στον κόσμο. Αρχίζω από τι παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ποιε είναι αυτές, περιορισμένοι πόροι, αυξανόμενο πληθυσμό. Αυτό ασκεί μεγάλη πίεση και στα τρόφιμα και στο κλίμα και στους φυσικούς πόρους. Τι βλέπουμε, ότι σιγά σιγά τελειώνει ε, η εποχή των ορυκτών καυσίμων και ενδεχομένω τώρα και τη πυρηνική ενέργεια με αυτά που γίνονται. Και η οικονομία που βασίζεται στη βιολογία ε, ήδη απογειώνεται. Έχουμε από σήμερα τα βιοκαύσιμα της επόμενης γενναίας. Όλο και περισσότερα είναι τα πρατήρια που δίνουν και βιοκαύσιμα. Τα πολιτικά εμπόδια έχουν μειωθεί. Υπάρχουν κάποια οικολογικά εμπόδια. Μέχρι την επόμενη γενιά θα έχουμε και βιοχημική βιομηχανία ε, για τα πλαστικά, ε, για τα χημικά και ακόμα και για τα ή Όπως σας είπα, στην Ευρώπη εκμεταλλευόμαστε τη γεωργία μας. Τα απόβλητα της γεωργίας είναι μοναδική ευκαιρία για καινοτομία στη γεωργία. Υπάρχουν οι λύσεις, οι βιοτεχνολογίες. Μπορούσαμε έτσι να επενδύσουμε στην αυριανή τεχνολογία και υποδομή θα μειώσουμε τα διοξίδια και τα αέρια του θερμοκηπίου, θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και θα αυξήσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια, τον εφοδιασμό. Και σιγά σιγά λοιπόν θα πρέπει να περνάμε προς μια οικονομία που βασίζεται στη βιολογία. Να σας πω τι είναι το βιοδιηλιστήριο. Τι είναι. Λοιπόν, βλέπουμε δεξιά τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, σήμερα, ε, αριστερά μάλλον ε, δημητριακά, και απόβλητα και δεξιά βλέπουμε τι παράγουμε και σε εμπορικό επίπεδο και στην επόμενη γενιά των βιοκαυσίμων. Στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία να αυξήσουμε όμως και τις εισρωές, όχι μόνο τις εκροές, ε, αστικά στερεά απόβλητα ας πούμε και ε, τελικά ε, χημικά χωρίς ορυκτά καύσιμα. Ε, θα πρέπει να αρχίσουμε, η καινοτομία θα μας οδηγήσει παρακάτω, αλλά η επόμενη γενιά είναι η πρώτη ε, που θα έχει μια πλήρη οικονομία βασισμένη στη βιολογία. Ευτυχώς δίνεται μεγάλη προσοχή σε αυτό. Ο ΣΑ ε, θεωρεί το 2030 το 2,7% του παγκοσμίου ΑΕΠ θα προέρχεται από την οικονομία αυτή. Ε, το WWF επίσης λέει ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε ένα με δυόμιση δις τόνους διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2003 και ε, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μου λέει ότι θα εξοικονομήσουμε ε, περίπου 23 ε, δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Προβλέπετε λοιπόν ένα ταξίδι προς μια οικονομία χαμηλή σε διοξίδιο του άνθρακα. Από πού αρχίζουν όλα αυτά, από τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της οικονομίας με τη βιοτεχνολογία στη βιομηχανία μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων, το κάνουμε ήδη από τώρα. Στη συνέχεια είναι η μετάβαση στα βιοκαύσιμα της επόμενης γενιάς. Σήμερα υπάρχει αυτή η τεχνολογία και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα εμπόδια που υπάρχουν είναι εμπόδια πολιτικά. Επίσης, επόμενη γενιά. Επόμενη. Η Bloomberg πρόσφατα δημοσίευσε μία έρευνα που ε, κοιτάει το μέλλον των αποβλήτων. 25% ας πούμε πάρουμε από τα σημερινά γεωργικά απόβλητα και τα χρησιμοποιήσουμε ε, ε, στα βιοκαύσιμα της επόμενης γενιάς μπορούμε να μειώσουμε κατά 62% και να αντικαταστήσουμε τη ε, χρησιμοποίηση και την κατανάλωση βενζίνης μέχρι το 2020, να δημιουργήσουμε μέχρι ένα εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης ε, και σε ε, περιοχές της υπαίθρου που δεν αντικαθίστανται από άλλες θέσεις απασχόλησης και μειώνουμε τις εκπομπές διοξυδίου του άνθρωπου. Επόμενο ορόσημο τα πετροχημικά, να τα αντικαταστήσουμε από βιολογικό υλικό. Δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί ακόμα βέβαια. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο και εκεί θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Και θα πρέπει να επικεντρωθούμε πολύ σε αυτό, διότι η Ευρώπη έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη βιοτεχνολογία αυτή παγκοσμίω και είναι ένα από του λίγου τομεί που μπορούμε να αντέξουμε στη σύγκριση με τι Ηνωμένε Πολιτείε και στον ανταγωνισμό. Ε, ας κινητοποιηθούμε προ τα εκεί. Ποιε οι μελλοντικέ προοπτικέ. Τώρα είμαστε στη δεύτερη γενιά και θα πάμε προ την τρίτη. Δεν χρειάζεται έρευνα. Υπάρχει η τεχνολογία. Πρέπει να την αναπτύξουμε. Και η τρίτη φάση είναι νέα βιοηλικά. Για να φτάσουμε στους στόχους για μείωση του διοξιδίου του άνθρακα και να μπορέσει και η γεωργία να συνεισφέρει και να μην ε, ε, είναι ε, απλώς καταναλωτής ε, και να απομιζά ενέργεια. Τα ανανεώσιμα χημικά είναι στα σπάργανα ακόμα. Θα πρέπει να ανταγωνίζονται και στη μέση και στην απόδοση δεν παίρνουν επιδοτήσεις και χρειάζεται ολόκληρη νέα υποδομή στην Ήπεθρο. Να σας αναφέρω μερικά από τα έργα που έχουμε εδώ, τα projects. Dupont, Danisco, Rocket και πολλοί όμως εργάζονται με ε, μεγάλες εταιρείες δισεκατομμυρίων επενδύσεις για να προχωρήσει αυτός ο δρόμος των βιοκαυσίμων. Αν θέλουμε όμως να προχωρήσουμε σε αυτό το όραμα και σε αυτή την οικονομία, πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να στρώνουμε τον δρόμο, να, να ε, φτιάχνουμε δίνηστήρια στην Ήπεθρο, γιατί η μεταφορά κοστίζει πολύ. πολύ. Και δεν ξέρω, με το 2050 ή μετά από 100 χρόνια, μπορεί να μην χρειαζόμαστε βιοκαύσιμα, αλλά μπορούν εκεί τα εργοστάσια να παράγουν άλλα πράγματα αν δεν χρειάζεται πια ενέργεια. Αυτό που ζητάμε λοιπόν είναι ε, πολιτική ηγεσία από την Ευρώπη. Να μην χάσουμε την ευκαιρία που έχουμε τώρα, αυτή την καλή κρίση που μας επιτρέπει να περάσουμε προς τα βιοκάψιμα να αναπτύξουμε πλήρως τα βιοκαύσιμα της επόμενης ε, γενεάς με περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νίλσεν πολύ σημαντικό ο τομέα αυτό σίγουρα. Γεωργική πολιτική μα ενδιαφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα. Πάντα, γιατί τώρα έχουμε και νομοθετική, ξέρετε, εξουσία με τη συνθήκη της Λισαβόνας μας έδωσαν και ε, για να ξεπεράσουμε και την κλιματική κρίση, αλλά να και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και να εξασφαλίσουμε το μέλλον αυτού του τομέα. Ποιος ζήτησε το λόγο? Η Λίνα Εκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αυτές οι ομιλίες. Έχω μια σύντομη ερώτηση προς τον κύριο Νίλσεν. Είστε πολύ ταπεινόφρον και δεν μας εξηγήσετε πώς μπορούν τα προϊόντα σας να συμβάλλουν στην ανάλυση του κύκλου ζωής της παραδοσιακής παραγωγής εθανόλης. Γιατί εξετάζουμε διαφορετικές γενναίες βιοκαυσίμων. Η δυνατότητα όμως χρήσης της βιοχημίας σε συνδυασμό με τα γεωρικά απόβλητα είναι τεράστια. Αυτό το δυναμικό είναι τεράστιο και όπως είπε και ο Πρόεδρος, αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και έχουμε διαπραγματεύσει για τη νέα κοινή γεωρική πολιτική. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον για όλους. Κύριε Λαμπερτιέ, για τη χαλιβουργία. Έχω δύο ερωτήσεις. Υπάρχει και ένας εσωτερικός γνώμονας σε ό,τι αφορά τους, ε, υψικαμί... τις υψικαμίνους. Θέλω όμως τη γνώμη σας για το δυναμικό. Γιατί οι καλύτερες υψικάμινοι, μερικοί τουλάχιστον βρίσκονται στην Ευρώπη, αλλά άλλες δεν έχουν τόσο καλές επιδόσεις. Άρα το δυναμικό βελτίωσή τους είναι μεγάλο. Συζητάμε ε, από κοινού μερικές φορές το σύστημα εμπορίας εκπομπών και την κατάσταση στη Χαλιβουργία. Μία εταιρεία στη Βόρεια Σουηδία έχει το 90% του, ε, της παραγωγής ε, σιδήρου και συμβάλλει κατά 40% στην ευρωπαϊκή μηχανή. Για τεχνικούς λόγους δεν εμπίπτουν στην ε, πρόταση benchmarking και το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σε αυτή τη συγκριτική αξιολόγηση να συμπεριλάβει όλες τις εταιρείες χαλιβουργίας, αλλά όχι αυτές που έχουν το Iron Ore. There is only one big company. Κι όμως αυτές είναι έξι εταιρείε, αλλά δεν συμμετέχουν στην συγκριτική αξιολόγηση παρόλο, παρόλο το μεγέθο τους. Άρα δεν εμπίπτουν στο σύστημα εμπορία εκπομπών. Αυτέ οι εταιρείε ε, εισάγουν όχι τόσο ποιοτικό χάλιβα από άλλες, εταιρείες, από άλλες έξω ε, κοινοτικές εταιρείες και προτιμούμε μερικές φορές να εισάγουν κακής ποιότητας ε, άνθρακα παρά να εισάγουν από την ΕΛΚΟ, την Σουηδική εταιρεία που έχει πολύ πιο ποιοτικό χάλιβα. Ίσα του χάσει. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Νίλσεν. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για τη βιοχημία και τα βιοκαύσιμα της επόμενης γενιάς που χρησιμοποιούν ως βάση τους τα γεωργικά απόβλητα. Είναι πραγματικά ε, συναρπαστικές αυτές οι ιδέες, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με τις τη χρήση της γης, γιατί με την πρώτη γενναία βιοκαυσίμων είχαμε πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη χρήση της, ε, του εδάφους. Ακόμη και χρησιμοποιούμε γεωργικά απόβλητα που δεν επηρεάζουν τη χρήση της καλλιεργήσιμης γης, αλλά ίσως έχουν ένα αντίκτυπο στο, στον άνθρακα ακριβώς επειδή είναι περιορισμένη η γεωργική υγιή στον πλανήτη, δεν θα πρέπει η παραγωγή βιοκαυσίμων να επηρεάζει να περιορίζει ακόμη περισσότερο την ε, χρήση της καλλιεργήσιμης γης. Ευχαριστώ. Έβαλα και εγώ το όνομά μου ε, στον κατάλογο των ομιλητών και προς τους δύο θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Το 2008 αποφασίσαμε θαύματα για το πακέτο, για τη τεχνολογία, για τη δέσμευση και αποθήκευση του ε, άνθρακα, τα βιοκαύσιμα, μπορώ να σας πω και από τη χώρα μου. Τεράστια συζήτηση γίνεται για τα ένζημα για το ε10 το καύσιμο που ο κόσμος δεν το αγοράζει. Ε, γιατί είναι πρόβλημα επικοινωνίας. Υπάρχει στα πρατήρια, αλλά δεν το προτιμούν οι καταναλωτές. Και πέρα από πολιτικά κόμματα είναι τεράστια η αντίδραση και η αντίσταση σε αυτή τη τεχνολογία. Έχουν δημιουργηθεί και πρωτοβουλίες πολιτών ε, τοπικά κοινοβούλια ψηφίζουν κατά του CCS, εμείς μιλάμε για την κλιματική κρίση, αλλά η αποδοχή στα κρατημέλη και μιλώ για τη δική μου χώρα, γιατί αυτή ξέρω, τη Γερμανία, έχουμε τεράστιο πρόβλημα να πείσουμε τον κόσμο. Εγώ φωνήβω όντω εν τη ερήμο, άντε και με μερικού συναδέλφου που είναι πεπισμένοι από αυτά τα πράγματα, αλλά ο κόσμο όχι. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί και να μας πείτε αν το έχετε λάβει υπόψη σας αυτό, εάν το γνωρίζετε και πώς επικοινωνεί κανείς ως βιομηχανία για αυτά τα πράγματα. Και το κάψιμο ε10 έχει ε, δείξει στη Γερμανία ότι ο ένας ρίχνει το φταίξιμο στον άλλον, τελικά όλοι μαζί στην πολιτική και τούμπαλιν. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου απαντήσετε σε αυτό. Και οι δύο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις ε, για τη χαλιβουργία. Καταρχήν ό,τι αφορά τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίω. Όντως, ορισμένα εργοστάσια στην Ευρώπη είναι διεθνούς φήμης και έχουν πολύ καλές επιδόσεις. Σε ό,τι αφορά τι άλλες χώρες, η Ιαπωνία και η Κορέα έχουν εφάμιλε ε, επιχειρήσει ε, με τις ευρωπαϊκές. Χώρε όπως η Κίνα και η Ινδία, 45% της παγκόσμιας ε, παραγωγής χαλιβουργίας ήταν η Κίνα για το 2010 και κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσει στο 50% την επόμενη διετία. Κάθε φορά που υπάρχει μεταφορά παραγωγής χάλιβα ή αύξηση παραγωγής χάλιβα στην Κίνα ή στην Ινδία, έχουμε πρόβλημα διαρροής άνθρακα, γιατί οι χώρες αυτές δεν έχουν τόσο καλές επιδόσεις ε, εξοικονόμησης ενέργειας με εμάς ό,τι αφορά την χρήση άνθρακα για την παραγωγή ενός τόνου χάλιβα. Υπάρχουν διαφορές τώρα και μεταξύ μας, μεταξύ των καλύτερων και των λιγότερο καλών. 20% είναι το χάσμα μεταξύ των 10 καλύτερων ευρωπαϊκών ε, χαλιβουργιών και των ε, λιγότερο καλών. Γι' αυτό και μίλησα για το τεράστιο δυναμικό πρόοδο που είναι της τάξης του 10% στην Ευρώπη προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των ε, καλών χαλιβουργιών και των λιγότερο καλών και να αυξηθεί προς, να αναβαθμιστεί προς τα πάνω το, η γενική εικόνα. Σε ό,τι αφορά τα σύμπικτα τώρα, τα pellets, όντως ε, τα Σουηδικά είναι πολύ, τα ευρωπαϊκά σύμπικτα είναι πολύ καλής ποιότητας. Βέβαια η αγορά σύμπικτων είναι παγκόσμια, οπότε όταν γίνεται η αγορά στη Σουηδία ή τα αγοράζουμε στη Βραζιλία, η τιμή είναι ίδια, γιατί η αγορά όπως σας είπα είναι παγκόσμια. Σε ό,τι αφορά το γενικό απολογισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και συμπερίληψη στην, στον υπολογισμό της παραγωγής διοξιδίου του άνθρακα για την κατασκευή συμπίκτων. Από τη στιγμή που τα σύμπικτα δεν επιβαρύνονται με το διοξείδιο του άνθρακα που χρειάστηκε για να παραχθούν, έχουμε μία διαφορά για την βιομηχανία που τα παρήγαγε, αλλά για τον πλανήτη δεν υπάρχει διαφορά γιατί σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, το συνολικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είτε περιλαμβάνεται η διοξίδα του άνθρακα στον υπολογισμό της παραγωγής των συμπίκτων, είτε όχι. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τώρα της νομοθεσίας για τις κλιματικές αλλαγές, εδώ η συζήτηση είναι ευρύτατη. Και από τη στιγμή που υπάρχει ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών, Σίγουρα οι σιδηρουργίες, οι χαλιβουργίες έχουν κάποια κίνητρα να σημειώσουν πρόοδο σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά δυστυχώς σήμερα και με τις εφιστάμενες τεχνολογίες ελάχιστη είναι η πρόοδος που γίνεται. Μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε βέβαια τις ε, επιχειρήσεις και τα εργοστάσια προς τις καλύτερες ε, από αποδόσεις και επιδόσεις με μια καλύτερη ανταλλαγή των πρακτικών και με τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών. Σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας δηλαδή των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, το σύστημα εμπορίας εκπομπών μετά το 2012 μας ζητά να επιδείξουμε πρόοδο προ το benchmark της τάξης του 10% σε σχέση με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Και από τεχνική άποψη σήμερα δεν έχουμε την τεχνική λύση για να υλοποιήσουμε αυτή την πρόοδο του 10%. Χρειαζόμαστε και άλλη καινοτομία για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των εγκαταστάσεων μας, των υποδομών μας. Ο δρόμος είναι μακρύς γιατί θα πρέπει να γίνουν πειράματα στα εργαστήρια καταρχήν, μετά πιλωτικά προγράμματα στις βιομηχανίες, τα πειραματικά προγράμματα και εφαρμογή στι βιομηχανίε και είναι χρονοβόρα η διαδικασία. Στο σχέδιο συνδέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα και το στη Γαλλία, στο Iron Scheme, καθέσαμε τον τοσχέτο το Φεβρουάριο, θα εξεταστεί στην Επιτροπή το Μάιο, θα έχουμε την απάντηση στις αρχές του 2012 και αν μας δοθεί άδεια, θα αρχίσει η εφαρμογή πριν τα τέλη του 2015. Δηλαδή η εκμετάλλευση θα αρχίσει το 2016. Χρειάζεται τουλάχιστον μια πενταετία για να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί το σύνολο της διαδικασίας. Οπότε ο παράγων χρόνος είναι πολύ σημαντικός σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Να αρχίσω από τη δική σας ερώτηση πρώτα. Για την επικοινωνία και την αποδοχή του πληθυσμού. Να βγάλω και τα ακουστικά μου για να μην μπερδεύομαι. Τα βιοκαύσιμα είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί πριν από πέντε χρόνια ήταν ο Μεσσίας, ε, ο Σωτήρας και ξαφνικά έγινε πολύ γρήγορα από ο τράγος αυτός ο κλάδος. Αυτό εξαρτάται από την αηφορία και τη βιωσιμότητα και έγινε και μεγάλη φασαρία βιοκαύσιμα απέναντι στα τρόφιμα. Μα τώρα πρόκειται για την επόμενη γενιά. Είναι το μέλλον, όχι μόνο για τις μεταφορές, αλλά και την κοινωνία που θα βασίζεται ε, στη βιολογία. Έχουμε καλά κριτήρια για την βιωσιμότητα και αυτό ισχύει για την επόμενη γενιά, γιατί η επόμενη γενιά δεν είναι επανάκια. Η βιομάζα είναι και αυτή ε, πεπερασμένη ε, πρώτη ύλη. Και μέσω μακροπρόθεσμα μία λύση έχουμε μόνο, βιοκαύσιμα. Βλέπουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αναπτύσσονται, αλλά αν θέλουμε ε, να προχωρήσουμε στο μέλλον ή είναι η λύση να είναι βιώσιμη η ε, οδός αυτή των βιοκαυσίμων και είμαστε ήδη στην επόμενη γενιά. Αλλά να μην μαζεύουμε πάρα πολλά απόβλητα, υπολείμματα από τη γεωργία, γιατί δεν θα πρέπει να ε, φτωχαίνει και το έδαφος. Θα πρέπει να, αφήνουμε ε, πρώτες ύλες να, να, ε, της Ιοργίας να εμπλουτίζουν το έδαφος, να μην το αποδυναμώνουμε. 25% ας πούμε κατά μέσο όρο, αυτό λένε οι πανεπιστημιακοί, ή μέχρι 50% αλλά αυτό και πάλι είναι δοκιμή η μελέτη που έχει γίνει, εξαρτάται πάρα πολύ ε, από την ποιότητα του εκάστοτε εδάφους. Πάντως είναι τεράστια η δυνατότητα που έχουμε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα υπολείμματα ε, σίτου στα χωράφια και ε, άλλων ε, καλλιεργειών για οργανικά στερεά απόβλητα. Υπάρχει δυνατότητα και θα πρέπει να μπορούν να διαφοροποιούν και τις πηγές εισοδήματός τους οι αγρότες. Θα πρέπει να ανεβαίνουμε εκεί στην αλυσίδα αξιών και στη δυνατότητα ενίσχυσης του εισοδήματος των αγροτών. Δεν υπάρχουν πανάκες λοιπόν και χρήστες λύσεις, αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία η επόμενη γενιά. Αλλά η επόμενη γενιά είναι επόμενη πενταετία, γιατί ο κόσμος δεν βλέπει τόσο μακριά ε, στο μέλλον. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα αυτή και θα πρέπει από τώρα να ε, δούμε και την οδηγία για τις ανανεώσιμες που λέει 10% για το 2020 να προέρχεται από ανανεώσιμες, αλλά το πλαίσιο για την επόμενη γενιά είναι πολύ ασθενές. Εάν δούμε τα εθνικά προγράμματα δράσης ε, των κρατών μελών που αναφέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ θα φτάσουν σε αυτό το στόχο, είναι πολύ μικρή η αναφορά για να μην πω ανύπαρκτη στην επόμενη γενναία. Υπάρχει μία πρόληψη για διπλή ε, προσμέτρηση, δηλαδή 5% πρώτα και αργότερα 5%. Αλλά για τους επενδυτές αυτό δεν ε, εξυπηρετεί. Είναι πολύ ακριβές οι πρώτες εγκαταστάσεις, τα πρώτα εργοστάσια. Και αυτή η διπλή, ε, ο διπλός υπολογισμός δεν δουλεύει. Δεν εξυπηρετεί. Αν θέλουμε όμως να προχωρήσουμε σε αυτό το όρεμα μιας οικονομίας που να βασίζεται στη βιολογία, χρειάζεται ειδική ε, πρόβλεψη, ε, έτσι ώστε ε, τα προϊόντα της επόμενης γενεάς να μπαίνουν στη βενζίνη και να κυκλοφορούν τα καύσιμα. Καλή η οδηγία. Επίσης η ενεργειακή, η φορολόγηση της ενέργειας. Ε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα γίνει η οικονομία μέχρι 90% στο διοξείδιο του άνθρακα από τα βιοκαύσιμα σε σύγκριση με τη βενζίνη. Και αυτό είναι επιχείρημα και φορολογικό και κόστος. Και πάλι όμως το κλειδί για την επόμενη γενιά είναι όχι άλλη έρευνα και ανάπτυξη. Έχουμε την έρευνα, έχουμε την ανάπτυξη, έχουμε την τεχνολογία, τα βιοδιελιστήρια. Ε, ξέρουμε τα εργοστήρια ζαχάρεως που παίρνουν την κυταρίνη και την κάνουν ζάχαρη. Ε, τώρα το πάμε ακόμα παραπέρα. Ε, και ε, η κοινωνία θα τα ζητάει αυτά και θα είναι τεράστια η ζήτηση στο μέλλον για τα βιοχημικά και αυτό το λένε πολλές μελέτες. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά χρειάζεται να δημιουργήσουμε τη ε, τεχνολογία για τα βιοκαύσιμα της επόμενης γενιάς με αηφορία, με βιωσιμότητα και να βρούμε ένα στόχο. Δεν ξέρω, 20%, 30% για μεταφορά, ε, για οδικές μεταφορές, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Αλλά υπάρχουν ε, στα χωράφια οι πρώτες ύλες, εκεί θα πρέπει να πάμε να τις βρούμε. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, ξέχασα να απαντήσω σε ένα τμήμα της δικής σας ερώτησης για την αποδοχή από το κοινό. Είναι σαφές ότι οι νέες μέθοδοι που αναπτύσσουμε βασίζονται όλες στη δέσμευση και αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα και αυτό είναι πρόβλημα αποδοχής σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να το λύσουμε αυτό, να το φροντίσουμε. Αυτό αφορά και τα 8 ε, σχέδια και τα οχτώ προγράμματα επίδειξης, ε, τουλάχιστον το ένα ε, δεν αναφέρεται στο CCS, τα υπόλοιπα όμως 7, ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα της αποδοχής από τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ωραίο αυτό το συμπέρασμα για το δεύτερο πάνελ. Για την έρευνα, η έρευνα και τα προϊόντα της θα πρέπει στο τέλος να γίνονται αποδεκτά μετά από επικοινωνία και ενημέρωση του κοινού. Και ερχόμαστε τώρα στο τρίτο πάνελ. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο μιλητές. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Ε, νέα η κλάδη παραγωγής, ε, βιοχημεία και βιομηχανία είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάντα στην Επιτροπή μας. Ερχόμαστε τώρα στο τρίτο πάνελ και παρακαλώ και τους δύο μιλητές να έρθουν εδώ. Παρακαλώ, περάστε. Για να προλάβουμε να τηρήσουμε λίγο το χρόνο μας και να έχουμε και τη δυνατότητα ε, ερωτήσεων. Έχουμε λοιπόν και καλώς ορίζω θερμότατα τον κύριο Κάρστε Νόιχοφ από το Ινστιτούτο ε, Οικονομικής Έρευνας του Βερολίνου και τον Τζέρεμι Νίκολσον που είναι διευθυντής από το Ηνωμένο Βασίλειο από τους εντατικούς χρήστες ενέργειας. Θα σας πω, έχετε το λόγο, παρακαλώ να τηρήσετε και το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε για την συζήτηση αυτού του μονίμως επίκαιρου θέματος. Τι έγινε το 2007 όταν εξετάζαμε την την εφαρμογή μια οδηγία και τον αντίκτυπο στη διαρροή άνθρακα. Όταν μιλούμε για τη διαρροή άνθρακα, δούμε τον ορισμό τη διαρροή του άνθρακα. Αυτό που μα ενδιαφέρει σε ό,τι αφορά τη διαρροή είναι ότι εφαρμόζουμε πολιτικέ σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο που δημιουργούν ενάυσματα ώστε οι εργασ... τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν πολύ άνθρακα για την παραγωγή τους να μεταφέρονται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Βέβαια, έχουν γίνει πολλές μετακαταστάσεις ε, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι κλιματικές αλλαγές που... Ε, οι κλιματικές πολιτικές που υιοθετούμε να μην πυροδοτούν αυτές τις αλλαγές. Γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ κακό παράδειγμα ε, για άλλες περιοχές του κόσμου. Να υιοθετούμε λοιπόν ένα καθεστώς μια πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη βιομηχανία θα πρέπει να δούμε τι αντιμετωπίζει ο βιομηχανικός κλάδος. Αν η κλιματική πολιτική οδηγεί σε υπερβολικό άχθος οικονομικό. Εμείς κάναμε την μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλες χώρες παράλληλα, παράλληλα παραδείγματα έχουμε. Αν έχουμε 20 ευρώ σε σχέση με τα κονδύλια που αναφέρονται. Βίδαμε 15 με 20 τομεί, όπου το κόστος, η αύξηση του κόστους ε, της κλιματικές πολιτικές είναι σημαντικό. Έχουμε καταρχήν στο μπλε την αύξηση του ηλεκτρισμού και το γκρι χρώμα ε, την αύξηση του κόστους αν χρειαστεί να αγοραστούν όλε αυτέ οι άδειε για να πληρωθεί η, η επιβάρηση από τον άνθρακα. Θα πρέπει επίση σε δεύτερη φάση να εξετάσουμε κατά πόσο, ποια ε, κατά πόσο υπάρχει αντίκτυπος στην, στην δραστηριότητα. Στην περίπτωση των διελιστερίων δεν έχει νόημα, δεν έχει διαφορά, γιατί τα διελιστήρια μπορούν απλώ να αυξήσουν τη δυνατότητά του. Δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν περισσότερα και οι αλλαγέ σε τελική ανάλυση δεν είναι μεγάλε. Παρ' όλα αυτά, στι πολιτικέ συζητήσει που γίνονται, οι βιομηχανίες και τα συνδικάτα αλλά και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ανησυχούν για τη διαρροή άνθρακα, κάτι που οδηγεί όμως σε, σε ένα πολύ γενικό ορισμό για το ποιες, ε, ε, ποιοι κλάδοι μπορούν να επηρεάζονται από τη διαρροή άνθρακα. Και τελικά κίνδυνος διαρροής άνθρακα υπάρχουν, υπάρχει και πολλές βιομηχανίες. Βέβαια, ε, οι περισσότερες από τις βιομηχανίες αυτές έχουν δωρεάν άδειες, Πόσες δωρεάν άδειε όμως λαμβάνουν οι βιομηχανίε ανάλογα με το κόστος που αντιμετωπίζουν και βλέπουμε το 2009 οι περισσότεροι τομεί λαμβάνουν περισσότερες άδειες ε, ε, δωρεάν από ότι η αύξηση του κόστου που είχαν, τουλάχιστον για το 2009. Το 2009 μάλιστα ήταν ε, και η αρχή της οικονομικής κρίσης. Στο 2010 έχουμε χειρότερα ακόμη αποτελέσματα, αλλά ακόμη και για το 2008, πριν την οικονομική κρίση, είδαμε ότι η Χαλιβουργία έλαβε 20% περισσότερες ε, δωρεάν από ότι είχε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Με την περιβαλλοντική μας πολιτική δηλαδή, εξασφαλίζουμε ε, τη... να μην αντιμετωπίσουν συμπληρωματικό κόστο οι βιομηχανίε που θα διατρέχαν κίνδυνο διαρροή άνθρακα. Επίσης, ό,τι αφορά την διαμόρφωση των συγκριτικών αξιολογήσεων, του benchmark, ας μην ασχοληθούμε με αυτό τώρα, γιατί ήταν πολύ τεταμένη συζήτηση. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να επενδύσουμε σε βιομηχανίες χαμηλής χρυσάθρακα και πώς θα γίνουμε ανταγωνιστικοί και σε αυτό το τομέα. Δεν νομίζω ότι υπήρξε διαρροή άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτία τη περιβαλλοντική πολιτική μάλλον επωφελήθηκαν στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οι βιομηχανίες από την πολιτική μας για τις κλιματικές αλλαγές. Δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε σημαντικό φαινόμενο διαρροής άνθρακα με την κατάσταση των επιχειρήσεων εξαιτία των κλιματικών μας και περιβαλλοντικών μας πολιτικών. Κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι τι γίνεται σε δύο δραστηριότητες, το χαλκό και το αλουμίνιο. Αυτές οι βιομηχανίες έχουν μόνο το άμεσο κόστος ε, από την αύξηση της τιμής του ηλεκτρισμού, αλλά όχι από το κόστος του διοξιδίου του άνθρακα, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, γιατί απλώς χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό. Είναι δύο τομείς που μπορούν να τύχουν και κρατικών επιχορηγήσεων και μάλιστα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για το τι κατευθυντήρες γραμμές πρέπει να ακολουθήσουν οι χώρες σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς όμως που ε, όταν είχαν πρόβλημα καλύφθηκαν από τις δωρεάν άδειε. Περισσότερο η αύξηση της τιμή του ηλεκτρισμού είναι πιο καθοριστική. Ο ανταγωνισμό επηρεάζει από διαφορετική άποψη. Χάσαμε δύο χρόνια στη συζήτηση για τη διαρροή του άνθρακα και δεν συζητήσαμε για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Εκεί άλλε χώρε ήταν πολύ πιο αποτελεσματικέ όπως φάνηκε και από το πενταετές ε, πρόγραμμα της Κίνας. Και στο παράρτημά μας στην Κίνα είδαμε τι έγινε με το προηγούμενο πενταετές πρόγραμμα που τελείωσε πέρυσι. Η Κίνα ε, δεσμεύτηκε να αυξήσει την ε, ένταση ενέργειας, να βελτιώσει την ένταση ενέργειας κατά 20% και υλοποίησε το στόχο της. Τώρα ο επόμενος στόχος της Κίνας για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης είναι 16% για την ένταση ενέργειας και 17% για την ε, ένταση άνθρακα. Κατά πάσα πιθανότητα θα υλοποιήσει το στόχο μέχρι το 2020 να μειώσει κατά 45 με 50% τη, τη χρήση άνθρακα. Η Κινέζικη κυβέρνηση υιοθέτησε διάφορα μέτρα. Βλέπετε εδώ οι πρώτες χίλιες ε, εταιρείε παραγωγής είναι αυτές που είχαν και τις καλύτερες αποδόσεις ε, σε ό,τι αφορά την ε, εξοικονόμηση. Και στο νέο πεντετές πλαίσιο η Κίνα θα αυξήσει τις δαπάνες στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη κατά 2,2% του ΕΠ προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί αλλά και να λάβουν υπόψη και ε, νέες τεχνολογίες που δεν χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι πώς να δημιουργήσουμε πρόσφορο περιβάλλον που θα είναι ελκυστικό για τους επενδυτές ε, αλλά και για τη χρήση ε, τεχνολογιών χαμηλής ενέργειας. Και μάλιστα ο οδικό χάρτης για το 2050 είναι ένα καλό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και όπως ακούσαμε και σήμερα το πρωί, ε, οι επιχειρηματίες χρειάζονται ένα σταθερό πλαίσιο να ξέρουν ε, τι θα γίνει στο μέλλον και να μπορούν να προβλέψουν τις συνέπειες από τις επενδύσεις τους. Ο, οδηγός, ο οδικός χάρτης του 2050 είναι αποτελεσματικός από αυτή την άποψη, αλλά θα, για να είναι αξιόπιστος θα, θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες πολιτικές και μάλιστα με δέσμευση των, πολιτικ, των κρατών ότι θα τις εφαρμόσουν. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε πολιτικές ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να δούμε και τι έκανε μέχρι στιγμή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών και μάλιστα με, μετά από ετήσια αξιολόγηση ε, που κάναμε, είμαι πολύ πιο αισιόδοξο για το σύστημα εμπορία εκπομπών και τα αποτελέσματά του για τρει λόγου. Αυτό το σύστημα στηρίζεται σε διαδικασίε λήψη αποφάσεων των εταιριών σε διάφορε διαστάσει. Αν δούμε πώ μια εταιρεία κάνει τι στρατηγικέ επιλογέ, καταρχήν θα πρέπει να τραβήξουμε την προσοχή τη διαχείριση, ε, να υπάρχει σαφήνιση ότι αφορά τι επενδυτικέ επιλογέ και μετά να έχουμε σωστό τρόπο εφαρμογή αυτών των επενδυτικών επιλογών. Πώ επηρεάζει το ETS σε ό,τι αφορά την απόσπαση προσοχή των εταιριών. Όλε οι εταιρείε με τι οποίε μιλήσαμε είπε ότι είναι σημαντική μακροπρόθεσμη στόχη, αλλά πολλέ φορέ συγκεντρώνονται συγκεκριμένα συστήματα ε, υποστήριξη τεχνολογία, αλλά και στο σύστημα εμπορία εκπομπών, ένα ιδιασμός. Επίση, αφήνει ω προ τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα της πορείας, ε, της εξέλιξης του ETS για τις εταιρείε. Μερικές φορές βέβαια η πορεία αυτή δεν ευθυγραμμίζεται με τους μακροπρόθεσμους στόχους ε, για το μείωση των εκπομπών ε, για την Ευρώπη. Επίσης, αν υπάρχει αντιστάθμιση το άνθρακα, θα πρέπει να επιταχυνθεί η μείωση των καψερίων. Κάτι όμως που είναι επισφαλές για τις επενδύσεις. Και άρα μακροπρόθεσμα θα γίνει το σύστημα πιο επαχθές για την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή, τη διευκόλυνση εφαρμογής σχεδίων ε, που δεν χρησιμοποιούν πολύ άνθρακα. Η τιμή του άνθρακα είναι σημαντικό, γιατί από σκοπιάς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από ε, πλευράς Ευρωπαϊκών χωρών θα πρέπει τη τιμή του άνθρακα να εντάσσεται στην διαδικασία παραγωγής. Είτε μιλούμε για σκυρόδεμα, ε, τσιμέντο και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να δώσουμε ενάψματα ότι με την αποτελεσματική χρήση του χάλιβα και με το συνδυασμό καινοτόμων προϊόντων θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και στο στόχο της ενεργειακής απόδοσης το ETS δεν είναι και πολύ περιοριστικό ή πολύ αυστηρό σύστημα. Ίσως στο μέλλον χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αυστηρότητα και αυτό μας φαίνει στο ερώτημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ένα μηχανισμό στήριξη τη τιμή ε, του άνθρακα εξαιτία των αδυναμιών που παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορία Εκπομπών. Αν δεν ενισχύσουμε όμως το ευρωπαϊκό ETS, τα κρατη μέρη θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν εθνικές πολιτικές. Και εδώ έχουμε τη, τα διάφορα μεγέθη ανάπτυξη εταιριών στο παρελθόν και βλέποντας και τις νέες χώρες μέλη μετά το 2006 είδαμε ότι είχαμε μεγάλη αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης Γι' αυτό μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δείχνει ότι η ένταξη στο κοινό σχέδιο είναι πολύ επωφελής για την οικονομική ανάπτυξη και η εναρμόνιση το ίδιο. Είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα να συνδυάσουμε τις κλιματικές και τις περιβαλλοντικές αλλαγές και να τις εφαρμόσουμε σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να το δούμε σε κοινοτικό επίπεδο. Εν κατακλείδη, σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες για τη διαρροή άνθρακα, έτυχαν εκτενούς ανάλυσης το 2008. Δεν νομίζω ότι η διαρροή άνθρακα θα δημιουργήσει πρόβλημα, ακόμη και γίνουν πιο αυστηροί οι στόχοι. Αντιμετωπίζουμε όμως τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αυτό είναι υγιές. Χωρίς α, ε, ε, διεθνή ανταγωνισμό δεν θα είχαν κάνει πρόοδο οι βιομηχανίες μας. Βέβαια θα πρέπει να δημιουργήσουμε πρόσφορα έδαφος για αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Γιατί άλλο να ε, εξαγγέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα και άλλο η Κινέζικη. Και η Κινέζικη κυβέρνηση είναι πιο αξιόπιστη όταν εξαγγέλει ένα πρόβλημα. Θα πρέπει την ίδια αξιοπιστία να την δείξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε και οικονομικά προβλήματα και κλιματικές ανησυχίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νόιχοφ. κοιτώ ε, δεξιά από τον κύριο Νίκολσον, ο οποίος με το ζόρι κρατιόταν στην καρέκλα του την ώρα που μιλούσατε και θα του δώσω το λόγο τώρα να αντιδράσει. Ε, και ενδιαφέρουσα συζήτηση στο τελευταίο πάνελ αυτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πριν κάνω τα σχόλια μου για τους κλάδους που χρησιμοποιούν εντατικά ενέργεια, πρέπει να σας πω ότι σέβομαι τις απόψεις του προελίσαντα, αλλά διαφωνώ στο βάθος για το μέγεθος της απειλής για την ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία. Να σας πω γιατί. Ε, αλουμίνιο, ε, βιομηχανικά φυσικά αέρια, βιομηχανικά αέρια, συγγνώμη, χημική βιομηχανία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι εντατικοί χρήστε ενέργειας με διεθνή ε, ιδιοκτησία και σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό είναι εκτεθειμένα τα εργοστάσια αυτά σε διεθνή ανταγωνισμό και στα γειτονικά κράτη της Ευρώπης και από αλλού. Και ε, η ανταγωνιστική απειλή ποια είναι. Δεν είναι ε, η Ευρώπη να ανταγωνίζεται αυτούς που θέλουν να εισάγουν προϊόντα στην Ευρώπη. Είναι και εξαγωγική και θα πρέπει να είναι ε, ανταγωνιστική εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς αγορές και θα πρέπει να κοιτάμε με δασμούς και άλλους τρόπους πώς μπορούν να αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα. Διαφωνώ βαθύτατα με την πρόταση να ξεπεράσουμε το 20% μετά το 2020. Πριν από λίγα χρόνια μόνο ε, συμφωνήθηκε. Δυστυχώς το διεθνές περιβάλλον δεν βοήθησε καθόλου και λυπούμαστε γι' αυτό. Σήμερα γνωρίζουμε ότι καμία αναπτυγμένη οικονομία δεν θέλει να ε, επιβάλλει εκτός της Ευρώπης τη βιομηχανία της ε, ε, ε, σε τέτοιους ε, φόρους και σε τέτοιες επιβαρύνσεις. Το ξέρουμε αυτό. Καμία αναπτυσσόμενη οικονομία δεν θέλει να δεσμευθεί με απόλυτους στόχους. Σχετικούς εντάξει, 8, 9, 10, αν αυξάνεται το χρόνο η οικονομία στην Κίνα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με ένα σχετικό στόχο, όχι μόνο απόλυτο αριθμό. Γι' αυτό ε, ε, το θέμα της διαρροής ε, του διοξιδίου του άνθρακα σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ό,τι στο παρελθόν. Επίσης διαφωνούμε βαθύτατα με αυτά που λένε ορισμένοι Ευρωπαίοι πολιτικοί ότι η πιο φιλόδοξη στόχοι είναι και πιο προσεκτικοί. Το αντίθετο όταν είναι μια μικρή οικονομία είναι πιο εύκολο να αφαιρέσει το διοξίδιο του άνθρακα. Όταν είναι μεγάλη είναι πιο δύσκολο. Και επειδή έχει συρρυκνωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία φαίνεται ότι είναι λιγότερο το κόστος επειδή έχει συρρυκνωθεί η οικονομία. Και αν είχε περιοριστεί εντελώς και ε, εκμηδενιστεί τελείωσε η βιομηχανία, δεν θα είχαμε και κανένα κόστο περιορισμού του διοξιδίου του άνθρακα. Μα δεν πάει έτσι. Ε, πριν από λίγο είδαμε κάποιε γραφικέ παραστάσει ε, που συνέκριναν ε, τι παραχωρήσει με την ζήτηση για διοξίδιο του άνθρακα. Αλλά αυτό ήταν σε περίοδους και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο τσιμέντο και στο χάλιβο πέσαμε ε, κατά 30 και 40% Βεβαίω. γιατί ε, η βιομηχανική παραγωγή κατέρευσε σε τρόπο που δεν είχε φανταστεί κανένα τουλάχιστον εγώ όσο ζω. Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν προβλήματα με τη χορήγηση αδειών ε, και δικαιωμάτων, ότι να κάνουμε έτσι έχει η ζωή. Δεν είναι αποτυχία της αγοράς. Η αγορά δείχνει ότι φτάνουμε ε, κατά λάθο τους στόχους μας λόγω της ύφεσης <laughs> όχι ότι έχουμε κάνει καμιά τρομερή προσπάθεια ενεργητική. Και κατά τα άλλα, οι τομείς που καταναλώνουν πολύ ενέργεια, όπως είναι ε, οι αλλουργίες, ε, βιομηχανίες οι χαλιβουργίες, είναι τμήμα ε, της αλυσίδας ε, παραγωγής και χρειάζεται ε, παροχή, προσφορά ε, το θέμα είναι η προσφορά θα γίνει από την ε, Ευρώπη ή θα την εισάγουμε. Αυτό που μας απασχολεί δεν είναι μόνο ε, πόσο κοστίζουν οι άδειες και, τα δικαιώματα, αλλά το σωρευμένο βάρος της κλιματικής πολιτικής, με άλλα λόγια, φορολογία, το ETS και το άμεσο κόστος και το έμεσο κόστος όμως από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας. Αυτό αφορά όλες τις βιομηχανίες που καταναλώνουν πολύ ηλεκτρικό ρεύμα. Ακόμα και αν δεν υπήρχε θέμα, ας πούμε για τα βιομηχανικά αέρια, την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα που είναι πολύ χαμηλή, ε, σίγουρα ε, ε, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με την αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ακούσαμε, το 100% του κόστους το μετακυλίουν εταιρείε παραγωγή ε, ε, ηλεκτρική ενέργεια και επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή. Και επιπλέον έχουμε και ε, επιδοτήσει ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Αν δεν ήταν τόσο ακριβό το σύστημα επιχορήγηση των ανανεώσιμων και τόσο ακριβή η φόρη ενέργεια, ενδεχομένως να ε, είχαμε αναλάβει αυτό το κόστος χωρίς προβλήματα ανταγωνισμού. Δυστυχώς όμως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και καμιά φορά μας λένε ότι αυτή η πολιτική από μόνη της, δηλαδή με ένα πιο σκληρό στόχο μέχρι το 2020 για τις εκπομπές, αυτός ο μόνος στόχος ε, ε, σου λένε δεν είναι μοιραίος για το εργοστάσιο. Εντάξει, μπορεί. Είναι σαν να σου λένε όταν σε πυροβολεί κάποιο, ε, φας μια σφαίρα μπορεί και να μην πεθάνει. Ναι, αλλά άμα ε, φας πολλά σκάγια και πολλές σφαίρες μπορεί και κάποια από αυτά να σκοτώσει. Ε, είναι, είπαμε, ισορρευτικό το πρόβλημα, είναι πολλοί οι παράγοντες. Ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά μπορεί να μην είναι θερατηφόρος, αλλά το σύνολο μας κάνει να καταραίουμε. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι ένα στοιχείο μόνο δεν θα σας πειράξει. Και επιπλέον αυτά τα θέματα των benchmarking, της αξιολόγησης, δεν έχουν λυθεί ούτε για το χάλιβα, ούτε για τίποτα άλλο. Φοβάμαι λοιπόν ότι δεν είναι σωστό αυτό που ακούστηκε, ότι λύθηκαν αυτά τα προβλήματα, δεν έχουν λυθεί. Το θέμα της αντιστάθμισης για τις ηλεκτροεντατικές βιομηχανίες παραμένει μεγάλο πρόβλημα. Εδώ πρόκειται για βιομηχανίες εξαγωγικές και επομένως η προστασία των εισαγωγών δεν λύνει αυτό το πρόβλημα θα έπρεπε να είχα μιλήσει και για το πρόσθετο κόστος της επιχορήγησης μη οικονομικών ή μη αποδοτικών μεθόδων. ή και ανασφαλών ανανεωσίμων όπως τη νεολική ενέργεια. Εδώ μιλάμε για υπολογισμούς από τη Βρετανική κυβέρνηση. 60 με 70% αύξηση των τιμών μέχρι το 2020 μισές από τις οποίες αυξήσεις θα οφείλονται στις επιχορηγήσεις των ανανεωσίμων. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε γιατί η Ευρώπη αυξάνει το κόστος χωρίς να υπάρχει επαρκής λόγος. η βιομηχανία θα μπορούσε ίσως να αντιμετωπίσει το πρόσθετο αυτό κόστος αν υπήρχε όντως ήδη μια αγορά πιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης των εκπομπών του διοξιδίου. Αυτή τη στιγμή η Ένωση υπονομεύει τον ίδιο της τον κανόνα της συναλλαγής των εκπομπών με πρόσθετα μέτρα που αυξάνουν την τιμή της εκπομπής. Ποιος θα αγοράσει λοιπόν αυτά τα δικαιώματα. Έτσι καταστρέφονται οι αγορές και είναι πολύ επικίνδυνες οι ιδέες αυτές. Λυπηρό είναι αυτό. Τώρα για τις διαρροές. Υπάρχει μια δοκιμή των δύο αυτών απόψεων, κατά πόσον έχει υπάρξει ή όχι διαρροή δηλαδή για να δούμε αν έχει υπάρξει. Δεν βλέπουμε τι διοξίδιο παράγεται κατά τη διαδικασία παραγωγής, αλλά στην κατανάλωση από τους Ευρωπαίους καταναλωτές και καταναλώτριες. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες οι εκπομπές που αφορούν την κατανάλωση των αγαθών έχουν αυξηθεί, δεν έχουν μειωθεί. Δεν έχουμε απανθρακοποιήσει την οικονομία μας, την έχουμε απλώς αναδιανύμει διαφορετικά. Όσοι θέλουν διανοητικά τίμια αντιμετώπιση λοιπόν πρέπει να το δουν αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους. Τέλος, διαφωνώ απολύτως με το ότι πρέπει να ξεπεραστούν οι στόχοι του 2020. Όχι, θα χειροτερέψουν τα πράγματα έτσι. Και τώρα για να καταλήξει. Μάλιστα. Μου άρεσε πολύ η τοποθέτησή σας. Και επίση αυτό που είπατε, ότι μπορεί ένα μόνο μέτρο να μην ε, σα καταδικάζει, αλλά είναι ένα σύνολο μέτρο, μια δέσμη μέτρων και διάφοροι παράγοντε δρούν επιβαρυντικά και ει βάρο κάποιων κλάδων και χρειάζεται συντονισμό. Και αυτό που έχει στα χέρια της Ευρωπαϊκή Ένωση το σύστημα εμπορίας εκπομπών δεν είναι η καλύτερη λύση, ίσως είναι η δεύτερη καλύτερη λύση. Έχουν και φόρους ορισμένες χώρες και χρειάζεται καλύτερο συντονισμό σε αυτή την περίπτωση. Πολύ ενδιαφέρον το πάνελ αυτό. Και ε, η Λένα Εκ φυσικά έχει ζητήσει το λόγο, μοναδική. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ καταρχήν και τη γραμματεία, το προσωπικό και όλους όσους συμμετείχαν ε, στη διοργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόασης. Ήταν από τις πιο σημαντικές και μεστές ε, ακροάσεις που πραγματικά έδωσαν τέτοιο πλουτογνώσεις που στην επταετία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σπάνια ε, είχα ζήσει. Και χαίρομαι που ήταν πολύ, που ήταν παρόντες και παρά την ένταση έγραφαν πήρε το δός και κρατούσαν σημειώσεις. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί έχουμε πολλές ε, σημαντικές πληροφορίες πια και χάρη σε όλη αυτή τη γνώση μπορούμε να καταλήξουμε σε αποφάσεις μετά την επικοδομητική συμβολή αυτών των πάνελ. Σε ό,τι αφορά τις τιμές ηλεκτρισμού και την ενεργειακή απόδοση, εδώ και 7 χρόνια είχα εντατικές επαφές με την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και αυτό που με συναρπάζει πάντοτε είναι πως κάποιες βιομηχανίες έντασης ενέργειας είναι, αυτές είναι μια ομάδα που χρησιμοποιεί τη νέα, τις νέες τεχνολογίες και που αξιοποιεί τις δυνατότητες για τη μείωση της χρήσης ενέργειας, της χρήσης του ηλεκτρισμού προκειμένου να ωφεληθούν και οι ιδιοκτήτες της εταιρείας και οι εργαζόμενοι αλλά και η κοινωνία γενικώ. Αλλά υπάρχει Απ' την άλλη πλευρά, ένας μεγάλος αριθμός εργοστασίων που απέρριψαν αυτές τις δυνατότητες, δεν επένδυσαν στις κατάλληλες τεχνολογίες για να εξοικονομήσουν ενέργεια και κρίμα γιατί υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια προσιτά που θα οδηγήσουν και σε αύξηση του κέρδους τους. Αναφερθήκατε στη Χαλιβουργία που είναι μια βιομηχανία έντασης ε, ενεργειακής, ε, έντασης ενέργειας. Χρησιμοποιεί και άνθρακα και είναι τεράστιο το φάσμα των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και να εξασφαλίσουμε αηφόρο ανάπτυξη. Και μπορούμε να κάνουμε και αξιολογήσεις συγκριτικές ε, για το ποιο σύστημα δουλεύει καλύτερα και Φάνηκε και από το σύστημα εμπορίας εκπομπών ότι το καλύτερο αποτέλεσμα το λαμβάνει η εταιρεία που είναι κοντά στις ανάγκες τη αγορά. Επειδή στις 12 πρέπει να ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σα. και χαίρομαι που αναμεταδόθηκε και απευθείας αυτή η δημόσια κρόση και πολλοί θα την παρακολούθησαν από τις οθόνες τους και ελπίζω να μας δώσετε τις διαφάνειες και τις ομιλίες σας ε, και γραπτός για να μπορέσουμε να τις μετελητήσουμε επισταμμένως. Ζητώ συγγνώμη Ματίας. Εσύ κάνεις πολύ καλή δουλειά που προσπαθείς να συμμαζεύεις τις ομιλίες και να τελειώσουμε εγκαίρως, αλλά είναι από τις βασικές συζητήσεις που πρόκειται να κάνουμε αυτό το θέμα ε, για το κλίμα και τους στόχους. Θα ήθελα να ρωτήσω ε, τον κύριο ε, Νόιχοφ, αν μπορεί να απαντήσει στον κύριο Νίκολσον για αυτή τον ισχυρισμό ε, ότι είναι πολλά τα εμπόδια και τα βάρη που πρέπει να επομιστεί και τη φορολογία και τα άλλα. Αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο για το σωρευτικό πλεονέκτημα, τα πλεονεκτήματα. Δωρεάν άδειε πήρατε και στην πρώτη και στη δεύτερη ε, φάση και βγάλατε και χρήματα. Ήταν πολύ κερδοφόρες οι φάσεις αυτές και αυτό το δείχνουν οι μελέτες όλες. Και στην επόμενη ε, φάση πάλι για την ένταση ενέργειας, για τον κλάδο αυτό, ε, είναι δωρεάν η ενέργεια. Ε, είναι δωρεάν οι άδειε. Άρα Σα κάνουν δώρο ένα γεύμα, γιατί καμιά φορά λέμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα ω γεύμα δωρεάν, κάποιο αντάλλαγμα θα θέλει πάντα να έχει. Λοιπόν, έχετε και πλεονεκτήματα. Μα είπατε για κάποια πράγματα που σα βαραίνουν, ενώ τα άλλα, τι να κάνουμε, είναι ε, πράγματα που έχει ζωή. Ενώ το άλλο είναι ένα πιστόλι που σα βάζουν στο κρόταφο. Ε, ε, στη ζωή όμω καλό είναι να ψάχνουμε συμβιβασμού. Γιατί δεν μπορείτε να αποκρούετε τα επιχειρήματα των δωρεάν ε, αδειών, ότι εντάξει τι να κάνουμε αυτά είναι μέσα από τη ζωή ενώ το άλλο είναι μειονέκτημα. Έχετε και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και χρειάζεται λίγο μια κοινή λογική ε, από όλε τις πλευρές. Δεν έχετε μόνο σωρευτικά ε, μειονεκτήματα, έχετε και σωρευτικά πλεονεκτήματα και είναι κρίμα που δεν τα αναφέρετε αυτά. Δεν έχει ρωτήσει κανένα άλλο τίποτα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα και στου δύο μιλητέ μα για να απαντήσουν. Mm. Ευχαριστώ. Δεν αναφέρθηκα στα συσσωρευτικά αποτελέσματα, γιατί αυτά δεν τα έχουν καταλάβει μερικέ φορέ οι βιομηχανίε. Όντω υπήρξε ένα δυναμικό τέτοιο κέρδους, μια δυνατότητα κέρδους, ιδιαίτερα στην παραγωγή ενέργεια και στην πρώτη φάση του συστήματος εμπορία εκπομπών ήμασταν αρκετά επικριτικοί, γιατί δεν ε, ήταν δυνατή η πρόσβαση στο δανεισμό, αλλά Δόθηκαν και κάποιες δωρεάν άδειες, αλλά ε, το πρόβλημα δεν θα πρέπει να υπήρξε, ε, υπήρξε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι εταιρείε παραγωγή ενέργεια μπορούσαν να μετακυλήσουν το κόστος ε, των αδειών στις, στους χρήστες. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν ο αρχικό στόχο ε, του συστήματο εμπορία εκπομπών και η ιδέα ότι η παραγωγή ενέργειας ή μεταπητικές ενέργειες ε, θα καρπώνονται τα ωφέλη ε, από το σύστημα εμπορίας εκπομπών και θα έχουν και κέρδος από πάνω. Αν όμως έχουμε τις άδειες σε μια μεγάλη περίοδο και αν αυτή είναι η μέθοδος υπολογισμού που χρησιμοποιείται, ίσως όντως παρουσιαστεί υπερβολική χορήγηση αδειών. Υπάρχει όμως εδώ ένας επιχειρηματικός κίνδυνος και αναφερθήκατε στις, ε, στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι για το έργο που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την προσπάθειά της να εντοπίσει, να, να βοηθήσει τις ε, βιομηχανίες, αλλά νομίζω ότι καθυστέρησε κάπως. Και προ τι να προσπαθούμε να ελκύσουμε επενδύσει στην Ευρώπη από άλλε περιοχέ του κόσμου, όταν υπάρχει ο κίνδυνο εδώ, το θέμα του κινδύνου. Γιατί η φάση 3 είναι σχετικά κοντά. Και σίγουρα θέλουμε επενδύσει, αλλά υπάρχει αβεβαιότητα. Πώ είναι δυνατό με τέτοια βέβαιο κλίμα να προσελκύσουμε επενδύσει. Γι' αυτό έχουμε διαρροή των επενδύσεων όχι επειδή υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά υπάρχει αβεβαιότητα για το αν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν μπορούμε λοιπόν να χρονοτριβούμε άλλο. Θα πρέπει να καλύψουμε αυτή την αβεβαιότητα, γιατί η αβεβαιότητα είναι που αποθεί τι επενδύσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακάρι να είχα μιλήσει περισσότερα για τα σωρευτικά αποτελέσματα, αλλά δυστυχώ η βιομηχανία δεν τα αντιλαμβάνεται αυτά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό δεν τα ανέφερα. Συμφωνώ πολύ τους. Όσο έχουμε ανασφάλεια δεν πρόκειται να προσελκύσουμε επενδύσεις. Και αν δεν είναι ισχυρό το πλαίσιο και σαφές για το που θέλουμε να πάμε, διατηρούμε τη μεγάλη ανασφάλεια. Διαφωνώ με αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, ότι ο στόχος όταν είναι πιο ε, αυστηρός, ε, αποθαρρύνει επενδύσεις. Είναι κερδοφόρα επένδυση αυτό. Ε, θα αποκομίσουν ωφέλη όσοι επενδύσουν. Τώρα για το συγκριτικό, το σωρευτικό πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, εγώ δεν το βλέπω. Γιατί υπάρχουν παντού εξαιρέσεις σε όλα αυτά τα σχήματα για εκείνους που έχουν ένταση ενέργειας και το γερμανικό, για τη συνδυασμένη παραγωγή ενέργειας και θερμότητας. Και εκεί ε, οι εντατικοί ε, χρήστες ενέργειας έχουν εξαιρέσεις. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει αυτό το θέμα της ε, σωρευτικής επιβάρυνσης. Τώρα, να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα της βιομηχανίας βεβαίως. Ναι, χρειαζόμαστε ένα φόρο. Οι εταιρείε είχαν μια τετραετία για να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους. Ε, αυτό νομίζω είναι ένας λογικός ορίζοντας. Μπορεί να, να διαφωνούν εταιρείε που θέλουν γρήγορα να αποσβαίνουν τις επενδύσεις τους και να βγάζουν κέρδη. Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω αξίζει τον κόπο. Αν κάνουμε κακή βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη, αν δεν ε, προωθούμε ένα καινοτόμο περιβάλλον, θα χάσουμε θέσει απασχόληση, θα χάσουμε βιομηχανίε και θα αυξηθούν οι εισαγωγέ. Αυτό έχει να κάνει με τα κίνητρα που είναι ακατάλληλα που δίνουμε πολλέ φορέ. Και υπονομεύουμε ε, τις νέες ε, θέσει απασχόληση και υπονομεύουμε και τη σαφήνεια και την ασφάλεια αλλά δεν ορίζεται έτσι η διαρροή διοξιδίου του άνθρακα από την έκθεση του IPCC. Γιατί χρειαζόμαστε σύστημα εμπορία εκπομπών λοιπόν είναι εντάξει ε, απλώς οι φόροι που επιβάλλουν κάποια ε, κράτη-μέλη η κρίση μας έδειξε ότι πρέπει να έχουμε μια τροχιά, να είμαστε στραμμένοι προς το μέλλον, να ξέρουμε πού θέλουμε να πηγαίνουμε και τι αξιοπιστία. Είναι ένας ωραίος μηχανισμός το ETS να μεταφραστούν οι στόχοι σε μελλοντική πολιτική. Δεν είναι πανάκι, αλλά είναι σημαντικό στοιχείο. Και καλό είναι να καλύπτεται η Ευρώπη, γιατί οι περισσότερες εταιρείες τις οποίες ε, μιλούμε ε, κοιτάνε τι γίνεται στην Ευρώπη. Ε, αν θέλουμε να επιβάλλουμε μόνο εθνικέ πολιτικέ και τίποτα άλλο, αυτέ μπορεί να λειτουργούν σε μεγάλε χώρε όπω η Γερμανία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αποδίδουν στι υπόλοιπε χώρε. Και με ενδιαφέρει και το τι γίνεται στι υπόλοιπε ευρωπαϊκές χώρες. Μια τελευταία συμπληρωματική ερώτηση. Ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Παράκληση σύντομα όμω. Στίβαν Δεχρότε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω ένα ερώτημα για το set aside. Οι βιομηχανίες με εντατική χρήση ενέργειας συζητούν την ιδέα αυτή εδώ και πολύ καιρό, αλλά πρέπει πριν το 2013 να αρχίσει να εφαρμόζεται, γιατί πρέπει να γίνει προοδευτικά. Επίσης προτείναμε η πληστηριασμοί που γίνονται για τις άδειε εκπομπών να οργανωθούν καλύτερα γιατί μπορεί αλλιώς να αυξήσουν τις τιμές. Μέχρι το 2013 οι δωρεάν επιτρεπόμενες εκπομπές πώς θα οργανωθούν. Μπορείτε να μας πείτε και γι' αυτό μερικά πράγματα. Με εκπλήσει η ερώτηση αυτή. Λέτε ότι θα χαρεί η βιομηχανία εάν δεν χρειαστεί να πληρώνει για τις εκπομπές. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά να μπορεί να δεχτεί η βιομηχανία υψηλότερες τιμές, όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ. Διότι το θέμα εδώ είναι η υπονόμευση της πίστης στην αγορά. Θα υπάρξει χειραγώγηση των τιμών στη φάση αυτή, αυτό λέω. Δυστυχώς το ETS ε, ε, αυτή την επίκριση πρέπει να αντιμετωπίσει. Ότι δεν στοχεύει καν σε κάποια τιμή στοχευμένη. Μιλάει μόνο για το επίπεδο των εκπομπών και αν οι τιμές τελικά που θα χρειαστεί να πληρωθούν είναι χαμηλότερες από ό,τι υπολόγιζαν, τόσο το χειρότερο. Εγώ νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο το οργανώνουν είναι κάτι το οποίο θα ζημιώσει όλη τη βιομηχανία. Και θα πάψουμε πλέον να υποστηρίζουμε αυτό το πρόγραμμα της διεθνούς ανταλλαγής αδειών εκπομπής. Γιατί δεν είναι πια αξιόπιστο το πρόγραμμα αυτό με τις χειραγωγήσεις αυτές ως προς τις τιμές. Ναι, σιγά σιγά στο τέλος τη ε, της ακρόασης. Πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συνεδρίαση και όπως είπε η συνάδελφο Λένα Εκ, ευρύτατη συζήτηση, κάλυψε πάρα πολλά θέματα και το θέμα δεν περιορίζεται στο 20%, στο 30% ή αν θα παίξουμε την κολοκυθιά και θα τα βρούμε στη μέση. Δεν είναι τόσο απλή η συζήτηση, είναι πολυεπίπεδη γιατί είναι και η βιομηχανία μας πολύ σχηδή στην Ευρώπη και πολύ επίπεδη και θα πρέπει να ε, κάνουμε προσπάθεια να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο ε, της προστασίας του κλίματος και φέρουμε και ευθύνη εμείς που είμαστε κλεγμένοι ευρωβουλευτές εδώ. Ε, προς ποια κατεύθυνση. Να εξασφαλίσουμε την ευημερία στην Ευρώπη, τις θέσεις απασχόλησης να μην χαθούν, αλλά έχουμε και μια άλλη ευθύνη δεν θα έλεγα τώρα για το σύνολο του πλανήτη, γιατί εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Αλλά για την Ευρώπη έχουμε ευθύνη. Για τις εκπομπές ε, στην Ευρώπη, για τους ρήπους που εκπέμπουμε εμείς, φταίμε εμείς. Και εμείς έχουμε αυτή την ευθύνη να κάνουμε και το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο. Η πρόκληση θα είναι μεγάλη, λοιπόν, τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, μήνες. Ε, η ακρόαση αυτή έγινε στην Επιτροπή μας εσκεμένα τώρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτά που μάθαμε σήμερα να τα κάνουμε τροπολογίες και κείμενα. Και σας ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ήσασταν παρόντες σήμερα, αλλά και εσάς, τους ομιλητές μας και εμπειρογνώμονες που ήρθατε να μας τα πείτε. Και σε σύντομο χρόνο μας δώσατε τη θεώρηση των ειδικών. Και όπως όλα στη ζωή, κάπου στη μέση βρίσκεται η αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ και τη Γραμματεία και τους διερμηνείς που μας επέτρεψαν να γίνει αυτή η συνεδρίαση. Ξέρω πάντα πόση δουλειά χρειάζεται η διοργάνωση μιας τέτοιας ακρόασης, άξιζε τον κόπο όμως και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και όσους μας παρακολούθησαν στο ίντερνετ, τηλεθεατές και ακροατές. Μην νομίζετε, πολλοί μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο και έχει την ευκαιρία κανείς να παρακολουθεί το τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς να έρχεται στις Βρυξέλλες με διερμηνία. Λοιπόν, ο Μπάς ε, ε, είναι εισηγητής αρμόδιος καθήλυν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής συντάξης νομοδότησης. Και κλείνοντα, ξαναλέω αυτό που είπα στην αρχή. Η έκθεση των Ιούνιο δεν είναι, θα εγκριθεί, είναι σημαντική και θα είναι πολύ σημαντικότερη αν είμαστε ενωμένοι στο Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε ένα αποτέλεσμα με μία ψήφο διαφορά. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ισχυρό και δυνατό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σίγουρα δεν θα είναι τελευταία κρόση για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε και μας ενημερώσατε Καλή επάνωδο!